Να ξεκινήσουμε παρακαλώ. Καλημέρα. Βλέπω ότι η σκιώδηση οι περισσότεροι είναι εδώ. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα που έχουμε να συζητήσουμε και είναι και άλλοι που ξέρω ότι θέλουν να μιλήσουν. κυρία Πρέντερκαστ ήταν στην Κροατία χθε θα μα πει τα σχετικά φαντάζομαι αργότερα. Και η κυρία Βαϊσκέρπε που είναι αναπληρωτρία αλλά είναι εδώ και είναι και στάκτερη αγνωμοδότης Επιτροπής Περιβάλλοντος που ψηφίζει στις 10. Θα προσπαθήσουμε να τα έχουμε λοιπόν ε, περαιώσει μέχρι τότε. Αρχικά να πω σε όλους uh, ότι αυτή η συνεδρίαση μεταδίδεται. Όποιος θέλει λοιπόν μπορεί να παρακολουθεί στο διαδίκτυο τη συνεδρίαση και είμαι βέβαιος ότι πολλοί από τις επαγγελματικέ οργανώσεις που ενδιαφέρονται θα παρακολουθούν τη συνεδρίασή μας. Και στην ιστοσελίδα μας μπορείτε όμως να παρακολουθήσετε τη συνεδρία και να βρείτε και τις πληροφορίες για τα διάφορα θέματα και να εγγραφείτε για να λαμβάνετε και το newsletter της Επιτροπής. Περνάμε λοιπόν στο πρώτο σημείο της μερικής διάταξης. Θα δώσω το λόγο στο σκληρά εργαζόμενο, στην σκληρά εργαζόμενη Μπερναντέτ Περνιού και αντιπρόεδρο της Επιτροπής μας, αλλά πρώτα απ' όλα τον κύριο Τίτσερ, τον ε, αρμόδιο και τομεάρχη της Κομισιόν. Θέλω να τον καλωσορίσω. Ξέρω ότι έχετε μελετήσει πολύ προσεκτικά όλες τις τροπολογίες και έτσι θα έχουμε την δυνατότητα να συζητήσουμε αυτές τις τροπολογίες. Η Μπερναντέτ βέβαια θα μας πει και τη δική της άποψη επ' αυτόν. Η κυρία Φάις Γκέρμπερ όμως θα πάρει πρώτο λόγο επειδή πρέπει να πάει προς είπα να ψηφίσει στις 10 και μετά η κυρία Λεγκρίκ. Ο κ. Μπουζόη. Θα έρθουν και κάποιοι άλλοι. Ο κ. Γκουστάφσον νομίζω από την Κουίν εδώ. Εγώ εκπροσωπώ την κυρία Μακλάρκιν. ο κύριος Βάπτα θέλει να λάβει το λόγο, κυρία Πρέντεγκαστ επίσης. Όλοι θέλουν το λόγο. Τέλο πάντων, έχουμε και τι ψηφοφορίε στι 10 όπω είπα, αλλά φαντάζομαι ότι έχουμε χρόνο μέχρι τότε να ακούσουμε όλου. Η Μπερναντέτ Φερνιό λοιπόν έχει πρώτο το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, ιδιαίτερα τους σκιώδεις εισηγητές, με τους οποίους συνεργαστήκαμε με πολύ ωραίο τρόπο. Εχθές το βράδυ Είχαμε την πρώτη συνάντηση, θα ακολουθήσουν και άλλες. Από την αρχή της εργασίας που διεκπερώνουμε από καιρό όσον αφορά τις επαγγελματικές ε, δεξιότητες, έχουμε δει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όσον αφορά το θέμα αυτό, καθότι υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης και βεβαίως ε, νέες ευκαιρίες ε, για την εσωτερική αγορά και για την ευημερία των πολιτών. Πάρα πολλές τροπολογίες έχουν υποβληθεί. Και βεβαίως με τον τρόπο αυτό θεωρώ ότι μπορούν να βρεθούν καλές συμβιβαστικές λύσεις. Παρ' όλα αυτά θα μας χρειαστεί ίσως λίγο περισσότερος χρόνος από ό,τι αρχικά είχαμε προβλέψει. Γι' αυτό και ζήτησα από τη Γραμματεία η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας να γίνει στις 10 ε, Ιανουαρίου. Ελπίζω ότι οι συντονιστές θα επιβεβαιώσουν αυτήν την ε, πρόταση καθότι υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των πολιτικών ομάδων, να κερδίσουμε λίγο χρόνο, να έχουμε στη διάθεσή μας λίγο περισσότερο χρόνο. Οι τροπολογίες ε, βεβαίως έχουν υποβληθεί σε κάποια πολύ συγκεκριμένα θέματα. Πρώτον, όσον αφορά την επαγγελματική κάρτα, είναι ένα θέμα το οποίο συζητείται εδώ και πολύ καιρό. Και βεβαίως ε, έχουν υποβληθεί πολλές τροπολογίες για το θέμα αυτό η ισχύς θα την αποφασίζει το κράτος υποδοχής. Βεβαίως, για κάποια επαγγέλματα που αναγνωρίζονται αυτόματα, είτε αυτά τα επαγγέλματα που ανήκουν στο γενικό καθεστώς και έχουν επιπτώσεις στο θέμα της δημόσιας υγείας, αυτό ισχύει ήδη. Πιστεύω λοιπόν ότι θα βρεθούν συμβιβαστικές λύσεις. Τώρα, όσον αφορά τα νέα πιλωτικά πρόγραμμα, αυτό, προγράμματα, αυτό μπορεί να μας καθυστερήσει πολύ, καθότι πρόκειται για μια ηλεκτρονική κάρτα προαιρετική, η οποία θα λειτουργήσει χάρη στο σύστημα IME. Με πολύ περιορισμένο κόστος εξάλλου. Επειδή υπάρχουν λοιπόν πολλές τροπολογίες όσον αφορά την ε, κατεξουσιοδότηση ε, πράξη. Η κάθε περίπτωση αίτησης αυτής της κάρτας θα πρέπει να ακολουθείται από μία διαβούλευση μίας επιτροπής εμπειρογνωμόνων εθνικών κάτι που εξάλλου ορίζεται και στην τροπολογία 86 του αρχικού μου κειμένου. Κάτι το οποίο διευκρινίζει, αν θέλετε, εδώ το σημείο αυτό. Είμαι υπέρ, επίσης, της ε, μη αναγνώρισης. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος να υπάρξει απάντηση, αντίδραση από μέρους των αρχών και βεβαίως περιορισμός των ε, προθεσμιών. Αυτή η Αυτή η σιωπηρή, η έμεση αναγνώριση είναι κάτι που μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα του σχεδίου. Θεωρώ επίσης ότι οι 170, 285 και 92 τροπολογίες, οι οποίες ορίζουν ότι οι χώρες που δεν ρυθμίζουν αυτά τα επαγγέλματα θα πρέπει τουλάχιστον να επαληθεύουν, να ελέγχουν τα πτυχία και τους τίτλους. Όσον αφορά την μερική πρόσβαση, εδώ υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία που προτείνει εδώ να εξαιρεθούν τα επαγγέλματα στον τομέα της υγείας, της δημόσιας ασφάλειας και κάποια επαγγέλματα που αναγνωρίζονται αυτόματα. Εγώ συμφωνώ και με αυτές τις προτάσεις, εδώ βεβαίως πιστεύω και θα το συζητήσουμε βεβαίως με τους εισηγητές, τους κοιόδης και άλλους συναδέλφους που ενδιαφέρονται. Παρόλο λοιπόν που πιστεύω ότι οι εθνικές αρχές θα πρέπει να μπορούν να ε, παρεκκλίνουν σε κάποιες περιπτώσεις, να υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις ε, που θα γίνονται βεβαίως αναπερίπτωση και με την δική τους ευθύνη. Και εδώ λοιπόν πιστεύω ότι μπορεί να βρεθεί μια ε, ικανοποιητική συμβιβαστική λύση. Όσον αφορά τις μαθητείες, τις πρακτικές. Και εδώ θα πρέπει να κοιτάξουμε το θέμα της αμοιβή. Ξέρω ότι μπορεί να υπάρξει εδώ κάποιο νομικό πρόβλημα, αλλά μετά από συζήτηση με τις νομικές υπηρεσίες πιστεύω ότι και εδώ μπορεί να βρεθεί μια ικανοποιητική και προσαρμοσμένη λύση. Στα κοινά πλαίσια κατάρτισης. Είμαι πεπισμένη ότι πρόκειται για κάτι που μπορεί να μας δώσει πάρα πολλές δυνατότητες. Είναι κάτι που το θεωρώ αναπόφευκτο. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει εδώ να υπάρξει περισσότερη ευελιξία και συμφωνώ με τις προτάσεις του κ. Ρουφό και Μπουσόη. Έλεγχος γλωσσικής ε, ε, εκμάθησης. Εδώ το θέμα αυτό θα έλεγα ότι δεν είναι εύκολο να εφαρμοστεί καθότι υπάρχει αρμοδιότητα των εθνικών αρχών θα πρέπει να δούμε βεβαίως στην πράξη πώς αυτό μπορεί να εφαρμοστεί. Και ξέρετε ότι πολλές φορές κάτι που θεωρητικά μας βρίσκει σύμφωνους στην πράξη μπορεί να προκύψουν πολλά προβλήματα. Ο σεβασμός καταρχήν όσον αφορά ε, την ασφάλεια των ασθενών. Και εδώ υπάρχουν έννοιες που θα πρέπει σαφώς να τις ε, ελέγξουμε περισσότερο. Η κυρία Μακλάρκιν και η κυρία Τούρινεν έχουν υποβάλει τροπολογίες που πλησιάζουν τις τροπολογίες μου 37 και 75 που είχαν προκαλέσει ανησυχίες. Ίσως λοιπόν και εδώ θα πρέπει να επανέλθουμε στο θέμα αυτό και να βρούμε κάποιες λύσεις που να εγγυούνται την ασφάλεια των ε, ε, ασθενών χωρίς βεβαίως να αμφισβητούνται τα δικαιώματα των ειδικών του κλάδου. Οι νοσηλεύτριες, οι νοσοκόμες. Δεν μπορώ να μην αναφέρω αυτό το θέμα και τις τομεακές ε, διευθετήσεις για κάποια επαγγέλματα. Για τις νοσηλεύτριες, εδώ πρέπει να βρεθεί ταχύτατα μία λύση, καθότι η Ρουμάνες και Πολωνέζες νοσηλεύτριες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα όσον αφορά την κατάρτιση, την γενική ε, σχολική κατάρτιση, ε, εκπαίδευση, 12 ετή. Και εδώ συνεχίζει να υπάρχει μια πολύ σημαντική δυσκολία, παρόλο που εδώ και κάποιες εβδομάδες ε, έχει προχωρήσει ο διάλογος και έχει εξελιχθεί το θέμα. Κοιτάω τον Ανδρέα και την κυρία Βίσμπεργκερ και ξέρω ότι εδώ ενδεχομένως να μην έχει ξεκαθαρίσει το θέμα αυτής της διπλής δυνατότητες που μπορεί να μας οδηγήσει σε ανισορροπίες και σε διακρίσεις. Κάποιες τροπολογίες των συναδέλφων του ΕΛΚ είναι πολύ ασαφείς και ελλειπή θα έλεγα όσον αφορά την εγγύηση ποιότητας. Και για άλλη μια φορά δεν αμφισβητούμε εδώ αυτό το διτό σύστημα κατάρτισης που σε πολλούς τομείς, σε πολλά επαγγέλματα έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά του. Θέλω απλώς να δούμε εάν για τις νοσηλεύτριες υπάρχει σήμερα αντιστοιχεία μεταξύ της πραγματικότητας αυτού του επαγγέλματος και αυτής της ε, διάταξης. Θα πρέπει να δούμε ποιο είναι αυτό το διτό σύστημα κατάρτισης με ένα γάρσιο τρόπο, τι προβλέπει αυτή η οδηγία και βεβαίως ε, όλα αυτά τα σημεία συνεχίζουν να μην είναι τόσο ξεκάθαρα. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να μακρηγορήσω περισσότερο, η συζήτηση θα είναι πολύ πιο χρήσιμη. Το θέμα επίσης των συμβολεογράφων μας έχει απασχολήσει, υπάρχει όμως νομίζω πλειοψηφία. Και η πρώτη συνάντηση που έγινε χτες με τους Σκιώδης πιστεύω ότι θα οδηγήσει στην υποστήριξη των κρατών μελών του Συμβουλίου προς συμφέρον των επαγγελματιών και των πολιτών της Ευρώπης. Επαναλαμβάνω, η πρώτη συνάντηση με τους Κιώδης έγινε χτες. Στις 21 Νοεμβρίου θα γίνει η δεύτερη για μια μισή ώρα στο Στρασβούργο. Τρίτη συνάντηση θα προγραμματιστεί την πρώτη ε, εβδομάδα του Ιανουαρίου και ελπίζω να μπορέσουμε να ψηφίσουμε στις 10 Ιανουαρίου. Σας ευχαριστώ πολύ και βεβαίως έχετε όλοι το λόγο. Well, thank you very much Σας ευχαριστώ πολύ Μπερναντέτ. Ήταν πολύ ξεκάθαρα τα όσα μας είπατε. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες, αλλά καλύψατε πολύ έδαφος. Σε ό,τι αφορά την αναθεωρημένη προθεσμία, είπατε ότι ε, θα πρέπει οι συντονιστέ να το σκεφτούν και να αποφασίσουν, αλλά νομίζω ότι τα επιχειρήματά σας ε, ήταν ε, πολύ ισχυρά και σίγουρα αυτό που θέλουμε και ως Επιτροπή είναι να έχουμε μια ισχυρή θέση που μπορεί να υποστηρίξει η πλειοψηφία της ομάδας, κάτι σημαντικό και για την επόμενη φάση των συζητήσεων. Χωρίς να μπορούμε να προδικάσουμε, αλλά νομίζω ότι μάλλον ε, θα γίνει αυτό που ζήτησες. Να δώσω λοιπόν τώρα το λόγο καταρχάς στην κυρία Βάισμπεργκερ, συντάκτρια γνωμοδότης, που πρέπει να φύγει, δεν φαντάζομαι να παρεξηγηθούν οι άλλοι σκιώδεις. Λοιπόν, επειδή πρέπει να φύγεις τόσο άλλος, φαντάζομαι θα είσαι σύντομη. Πες μας λοιπόν ποια είναι η θέση σου και πώς ε, εξελίσσεται η κατάσταση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για την κατανόηση που ε, δείχνετε. Θα περιοριστώ στα πολύ ουσιαστικά σημεία. Υπάρχει μεγάλη συμφωνία σε πολλά από τα σημεία και πραγματικά θεωρώ ότι θα πετύχουμε ένα πολύ καλό ε, κείμενο, συμφωνία θα βρεθεί για τα επαγγέλματα στον τομέα της υγείας, ε, για τα δικαιώματα των ασθενών, την πρόσβαση των ασθενών, το θέμα της γλώσσας. Ναι, βεβαίω. Θέλουμε ένα υψηλό επίπεδο, ιδιαίτερα για τον τομέα τη υγεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ε, αρκετή γλωσσική, αν θέλετε, εκμάθηση, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα Για όλα λοιπόν τα θέματα που αφορούν τον τομέα της υγείας συμφωνούμε και είναι και ουσιαστικό αν θέλετε ε, σημείο αυτής της πρότασης. Περισσότερη κινητικότητα και εδώ συμφωνούμε γιατί θεωρούμε ότι θα γίνει ένα πολύ σημαντικό ποιοτικό βήμα ε, στην ενιαία αγορά. Το θέμα των νοσοκόμων, των νοσηλευτριών. Εδώ και θα πρέπει να κοιτάξουμε τις θέσεις ε, στο Συμβούλιο, αυτό δεν είναι μόνο γερμανικό αν θέλετε θέμα. Και η Ουγγαρία, ε, Σλοβακία, Λουξεμβούργο, Αυστρία έχουν μία θέση που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα όσον αφορά αυτήν την ε, οδηγία. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την εξαιρετικά ευχάριστη ατμόσφαιρα στην οποία διεκπεραιώνονται οι συζητήσεις μέχρι τώρα. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια, την κυρία Βερνιό, ε, για το θέμα βεβαίως ε, της ε, υγείας και ιδιαίτερα για τις νοσηλεύτριες. Την τελευταία φορά σας βρήκα πολύ πιο ανοιχτή και θα ήθελα πραγματικά να σας ευχαριστήσω. Πιστεύω ότι μπορούμε να ε, προοδεύσουμε. Το θέμα της δωδεκαετούς κατάρτισης. Μέχρι τώρα ξέρετε ότι οι θέσεις ε, δίστανται και εμείς έχουμε αυτό το σύστημα, το λεγόμενο βασικό εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο δίνει πρόσβαση σε, κάποιες, ε, σε κάποιους τομείς. Και εμείς είδαμε, παραδείγματο χάρη, ότι με το δικό μας σύστημα και με την πρόσβαση σε κάποιες επαγγελματικές καταρτήσεις μετά από μια συγκεκριμένη περίοδο ε, σχολικής ε, εκπαίδευσης, μειώσαμε σημαντικά την ανεργία των νέων. Έχουμε δηλαδή πολύ απτές και συγκεκριμένες επιτυχίες. Θεωρούμε ότι είναι λάθος δομικό διάρθρωσης και ότι δεν βελτιώνουμε την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης αν δεν αντιμετωπίσουμε το θέμα της επαγγελματικής κατάρτασης. Θα πρέπει εδώ αυτό που έχει γίνει σε εμά από το 77 να αρχίσει να αντιμετωπίζεται. Δεν μπορούμε να περιοριζόμαστε μόνο στο θέμα ε, της σχολικής εκπαίδευσης, ε, κατάρτισης. Δεν είναι αυτό, αν θέλετε, εγγύηση για την ε, ποιότητα μιας νοσοκόμας. Το να έχει πτυχίο μπακαλωρεά ή αμπιτούρ, αυτό δεν είναι προϋπόθεση για μία νοσοκόμα και το πόσο καλή θα είναι. Υπάρχουν και πολλά άλλα θέματα, ε, η εμπειρία, η οποία μπορεί να οδηγήσουν έναν εργοδότη να την επιλέξει. Και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θέτουμε απαιτήσει στις νοσοκόμες οι οποίες ε, δεν είναι οι σωστές. Παραδείγματος χάρη, ε, το θέμα της κινητικότητας. Ε, υπάρχουν πάρα πολλές νοσηλεύτερες που θα ήθελαν να φύγουν και να εργαστούν σε μια άλλη χώρα και εδώ υπάρχει το θέμα της αναγνώρισης των δεξιοτήτων και των προσώπων. Ο κύριος Φαπ και εγώ σαφώς και θα κάνουμε κάποια βήματα. Σήμερα στην ε, πρότασή μας θα είναι του, τουλάχιστον δεκαετής κατάρτιση. Συμφωνούμε λοιπόν για το διτό, αν θέλετε, σύστημα κατάρτισης. Αυτή όμως η δωδεκαετής με τον τρόπο που, απέτηση, με τον τρόπο που καθορίζεται, που ορίζεται και τα βήματα τα οποία εδώ φαίνεται να έχει κάνει η άλλη πλευρά για μας θα πρέπει να επανεξεταστούν. Ναι, βλέπουμε ότι εδώ είναι η τουλάχιστον δεκαετής κατάρτιση, αλλά και εδώ θα πρέπει να δείξετε λίγο περισσότερο, αν θέλετε, πνεύμα διαλόγου. Για μας το καθοριστικό σημείο είναι ότι από τη μία προτείνεται είτε 12 ετή κατάρτιση σχολική, είτε 10 χρόνια συν 3. Τελικά όμως, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αυτή η νοσοκόμα, αυτή η νοσηλεύτρια να μπορεί στο τέλος της κατάρτισής της να έχει τα απαραίτητα προσόντα για να μπορέσει να εργαστεί με ικανοποιητικό τρόπο. Ελπίζω λοιπόν να το δούμε έτσι το θέμα. Ελπίζω να μπορέσουμε σύντομα να μιλήσουμε για μια κοινή ε, συμβιβαστική λύση για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να φύγεις. Θα καλύψω αργότερα, Μπεναντέ. Τι θες να πεις τώρα κάτι. Πριν φύγει η κυρία Βαϊσκέμπη. Ναι, πάρα πολύ σύντομα, γιατί τα έχουμε ξανασυζητήσει πριν την ε, πράσινη εβδομάδα. Πράγματι, βλέποντας ε, τον κατάλογο των ε, ικανοτήτων, ε, είπατε κι εσείς ότι το παράρτημα είναι από το 77. Από το 77 μέχρι το 2012 σίγουρα οι ευθύνες, αρμοδιότητες των νοσηλευτριών, οι θεραπευτικές η επιστήμη, τεχνολογία έχουν εξελιχθεί. Και έχει αλλάξει και η δουλειά των νοσηλευτριών. και σίγουρα πρέπει αυτά να τα λάβουμε υπόψη. αλήθεια είναι λοιπόν. Προσοχή όμως, δεν είπα πριν ότι δεν το χρειαζόμαστε αυτό το διτό, γιατί μπορούμε να το βάλουμε εγκάρσια στην οδηγία, επειδή έχει δείξει ότι είναι θετικό σε άλλα επαγγέλματα. Οι νοσηλεύτριε είναι ένα επάγγελμα υγεία, πολύ σημαντικό και νομίζω ότι πρέπει να επανακαθορίσουμε τα κριτήρια, τα σχήματα και να έχουμε κάποιου ορισμού για να έχουμε όσο το δυνατόν μια εναρμόνιση προ τα άνω. Και βέβαια να μην κάνουμε διακρίσει. Όπω είπα, υπάρχουν νοσηλεύτριε που δεν γίνονται δεκτέ σε άλλε χώρε ήδη. Και αυτό είναι κακό και για την κινητικότητα. Πρέπει όμως να ε, βρούμε τη συμβιβαστική πρόταση που θα μας επιτρέψει να κάνουμε την ε, εναρμόνιση προς τα πάνω. Γι' αυτό ζήτησα περισσότερο χρόνο, επειδή είναι ένα σημείο τριβής ε, από την αρχή των συζήτησεων προσκρούμε σε αυτό. Πρόεδρος, πολύ καλά. Θα δούμε και τι θα γίνει και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος με Ευχαριστούμε την κυρία Βάση Γκέπρι για την πολύ καλή δουλειά. Περνάμε τώρα στους Σκιώδης. Λεγκρίπ, Πουσόη, Ρούλε, που την κυρία Τούρεν. Νομίζω εγώ θα εκπροσωπήσω την κυρία Μακλάρ και ο κύριος Γκούσταυσον. Α, δεν είναι εδώ ο κύριο Γκούσταυσον ακόμη. Τέλο πάντων. Και μετά Σφα, Πρέντεγκαστ, Κοράτσα, Μπίλτ, Κοράτσμαν, Σαλντεμόζε. Θα δούμε με το χρόνο πώ θα τα πάμε. Παρακαλώ λοιπόν να είστε όλοι σύντομοι. Είστε και εσεί στη λίστα. Μα σα διάβασα το όνομά σας το είπα. Λοιπόν, κυρία Λεγκρίπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι νομίζω ότι μπορούμε πράγματι να μας δώσουμε λίγο περισσότερο χρόνο, να αφαιρώσουμε λοιπόν λίγο περισσότερο χρόνο από τον προβλεπόμενο σε μία από τις 12 προτεραιότητες της πράξης για την νέα αγορά, έναν, σε έναν από τους 12 μοχλούς για την ανάπτυξη, όπως τους όρισε αρμόδιος για το θέμα επίτροπος. Νομίζω ότι είναι απόλυτα δικαιολογημένο να αφιερώσουμε λίγο περισσότερο χρόνο, λίγο περισσότερη δουλειά. Προσωπικά λοιπόν συμφωνώ και φαντάζομαι ότι θα το επιβεβαιώσουμε ότι δηλαδή θα αναβληθεί η ψηφοφορία της εκθέσεως της κυρίας Βερνιό στην Επιτροπή μας και θα ψηφιστεί τελικά στις 10 Ιανουαρίου κάτι που θα μας δώσει περισσότερο χρόνο για να φτάσουμε σε ισορροπημένες αποδεκτές συμβιβαστικές ε, προτάσεις τουλάχιστον από την πλειοψηφία των μελών αποδεκτές. Σήμερα, η ανταλλαγή απόψεων που έχουμε αφορά την πρώτη εξέταση περί των 600 τροπολογιών που έχουν κατατεθεί. Πρέπει να σας πω καταρχάς ότι η ομάδα μας ε, ε, είναι προσιλωμένη σε κάποιες εμβληματικές ε, από τις πρωτοβουλίες κομισιών και ε, των σχετικών τροπολογιών. Ε, θα σας αναφέρω κάποιες από αυτές. Φυσικά υπάρχουν πολλές και διάφορες απόψεις και στη δική μου ομάδα για κάποια ζητήματα, αλλά συνολικά υπάρχουν κάποιες ε, γενικές γραμμές. Πρώτα απ' όλα η Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Κάρτα, το έχω ξαναπεί και σε προηγούμενες ανταλλαγές απόψεων, δεν θα ήταν κατά την άποψή μου λογικό να επιμηκύνουμε τις προθεσμίες, υπάρχουν πολλές τροπολογίες ε, και κάθε μία προτείνει κάποιο άλλο νούμερο. Πρέπει να βρούμε μια λογική ε, συμβιβαστική λοιπόν λύση χωρίς να απομακρυνθούμε πολύ από τον ε, πρώτο στόχο, δηλαδή να έχουμε ένα συγκεκριμένο εργαλείο, καινοτόμο εργαλείο, αυτή την Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Κάρτα που τόσο την περιμένουν οι επαγγελματίε του κλάδου, αλλά και πολλοί βέβαια από του συμπολίτε μα. Σε ό,τι αφορά τη σιωπηρή αναγνώριση, όπω το είπατε και εσεί, κυρία Συγήτρια, και για αυτό το θέμα υπήρξαν πολλά σχόλια και κατατέθηκαν σχετικά πολλές τροπολογίες. Πιστεύω ότι αυτή η σιωπηρή έγκριση, ε, αναγνώριση πρέπει να διατηρηθεί. Πρόκειται για μια αρχή και για μια πρακτική που πηγαίνει προς την κατεύθυνση που εμείς επιθυμούμε για τη διευκόλυνση, την απλοποίηση, την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα για τη δημιουργία μιας πραγματικά ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας ε, που θα αξίζει να φέρει αυτό το όνομα. Σίγουρα περίπλοκες ε, θα είναι συζητήσει για το θέμα αυτό σε άλλα θεσμικά όργανα. Το βλέπουμε ήδη στο Συμβούλιο, ιδίω εκεί το βλέπουμε. Πρέπει λοιπόν να έχουμε υπόψη μας ότι έχουμε περιθώρια λιγμών και διαπραγματεύσεων και καλό θα ήταν να παραμείνουν ανοιχτά αυτά τα περιθώρια ως το δυνατόν περισσότερο. Και βέβαια και η αρχή της οποία αναγνώρισης και αποδοχής ξέρουμε ότι υπάρχει σε ό,τι αφορά την ελευθερή παροχή υπηρεσιών. Και εμείς οι ευρωβουλευτές νομίζω πρέπει να επαγρυπνούμε και να μην ε, χάσουμε αυτή την αρχή της οπήρης αναγνώσης. Τώρα, για να είμαστε και ισορροπημένοι, θα ήθελα να έχουμε μία αναστολή των προθεσμιών ε, δύο εβδομάδων σε περίπτωση που χρειάζεται συμπληρωματική ενημέρωση που να ζητηθεί από ένα κράτος μέλος για τα επαγγέλματα του τομέα της υγείας να έχουμε μια αναστολή των προθεσμιών για να μην υπάρχουν καταχρήσεις. Και όταν υπάρχει ρητό αίτημα για παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών. Νομίζω θα μπορούσαμε να εξετάσουμε τότε το ενδεχόμενο αυτό. Όταν το κράτος ε, ε, έχει λάβει έτοιμα να παράσχει συμπληρωματικέ προφορίε μέσα σε μια εβδομάδα. Σε ό,τι αφορά τα κέντρα παροχή βοήθεια, ναι, μεν θα πρέπει να συμμετέχουν και στην προετοιμασία των φακέλων και να μπορούν οι επαγγελματίε ε, να έχουν επαφή, αλλά όχι όμως ε, να εξουσιοδοτηθούν ή να επιφορτιστούν με την χορήγηση της Ευρωπαϊκής Επαγγελματικής Κάρτας. Τέλος, συμφωνώ και θέλω να αναφερθώ και στα επιχειρήματα της συναδέλφου της κυρίας Κοράτσα Μπίλτ και της κυρίας Πέλτς, πάντα για την επαγγελματική κάρτα. Νομίζω πρέπει να προσέξουμε για να μην ε, τελικά δημιουργήσουμε ένα εργαλείο, όπως ανέφερε και η συγκήτρια, που θα είναι αντίθετο με τις πρακτικές που ισχύουν σε ορισμένες χώρες, όπου έχουμε ε, λίγα αριθμισμένα επαγγέλματα. Η Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Κάρτα πιστεύω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως ένα εργαλείο αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων σε ένα άλλο κράτος μέλο. και όχι σαν ένα μέσο να ρυθμίσουμε έστω και, και καλυμμένα τα απαιτούμενα προσόντα για ένα επάγγελμα μέσα σε ένα κράτος μέλος που όμως εκεί δεν ρυθμίζεται το συγκεκριμένο επάγγελμα και θα πρέπει να συμφωνήσουμε πάνω σε αυτό το σημείο και να φροντίσουμε να ληφθούν υπόψη οι σχετικέ τροπολογίε. Μερική πρόσβαση. Και εδώ υπάρχουν πολλέ τροπολογίε και εγώ έχω συντάξει αρκετέ σε ό,τι αφορά την μερική πρόσβαση που πιστεύω ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι πρέπει να βασίζεται σε ένα πραγματικό αίτημα το οποίο θα εξετάζεται, άρα θα περιορίζεται και κατά περίπτωση. Η μερική πρόσβαση πρέπει να παραμείνει όμως εξαίρεση και προτείνω μάλιστα εξαίρεση από τη μερική πρόσβαση όσων ε, είναι ήδη δικαιούχοι του συστήματος ε, αυτόματης αναγνώρισης. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση, μιλάμε το επάγγελμα των συμβολεογράφων, για να έρθω σε αυτό το εξέχον επάγγελμα. Για τη μερική πρόσβαση, λοιπόν, σε ορισμένες από τις αρμοδιότητες που ασκούν οι επαγγελματίες ε, αυτοί, είναι ένα θέμα το οποίο έθεσαν αρκετοί συνάλλευοι της Επιτροπής με τους. Δεν νομίζω ότι η οδηγία ε, έχει ως στόχο να εξαιρέσει ρητός αυτή στη, αυτά, την πρόσβαση σε, στο ένα ή στο άλλο επάγγελμα. Συμφωνώ λοιπόν με την εισηγήτρια. Και δεν είμαι υπέρ τη συμπερίληψη των συμβολιογράφων στο πεδίο εφαρμογή τη οδηγία αυτή χωρίς όμως να φτάσουμε και στο σημείο να αναφέρουμε εγγράφος και άρα ε, δεσμευτικά τη ρητή εξαίρεση των συμβολογράφων από το πεδίο εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Μια τέτοια ρητή μνήα θα ότι θα ήταν ατυχής, άστοχη. Επίσης νομίζω ότι σχεδόν όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να διατηρηθεί. Και σε ό,τι αφορά τις πρακτικές, θα πρέπει να δούμε τον ορισμό, αλλά δεν φτάνουμε βέβαια στο αν θα είναι ε, άμυστη ή ε, έμυστη ή ασκούμενη. Για την Επιτροπή Περιβάλλοντος και Υγείας θα δούμε τι θα γίνει. Έρχομαι στις νοσηλεύτριες. Στην ομάδα μου πολλοί έδειξαν και μια επικοδομητική στάση, πολύ ευφυή, εφάνταστη και δημιουργική. Καταθέσαμε μια τροπολογία που λαμβάνει υπόψη τον ε, σύστημα αυτής της διετής κατάρτισης, το οποίο όπως είπα αφορά πολλά κράτη, όχι μόνο την Γερμανία, αλλά και τη Γερμανία περιλαμβάνει. Όπως είπε και η συγγήτρια κυρία Βερνιό, πρέπει να προσέξουμε αυτό το σύστημα της διπλής εντοσαγωγικών αγωγικών αναγνώρισης να μην οδηγήσει τελικά σε διακρίσεις ε, και βλάψει ε, νοσηλεύτες οι οποίες θέλουν να μεταβούν στο εξωτερικό για να εργαστούν εκεί. Πρέπει πάντως να γίνει ένα πρώτο βήμα προς ε, έναν συμβιβασμό αυτό είναι η τροπολογία που έχουμε καταθέσει και ίσως αν αφιερώσουμε λίγη παραπάνω προσπάθεια και λίγο παραπάνω χρόνο θα βρούμε ίσως και μία άλλη ε, λύση ε, επεξεργαζόμενη μία κοινή συμμεβαστική τροπολογία. Η αναγνώριση τώρα αυτών των συστημάτων απλής αναγνώρισης που ισχύει σε πολλά κράτη. Ναι, είναι σίγουρα εθνικό θέμα, ε, υπάρχει εθνική αρμοδιότητα, αλλά όμως πρέπει να ληφθεί υπόψη το τι ισχύει σε κάποια κράτη. Στο πλαίσιο της αναθεωρημένης αυτής οδηγίας, δεν θα μακρηγορήσω άλλο, έθιξα αρκετά ζητήματα, χαίρομαι γιατί υπάρχει σχέ... μεγάλο πνεύμα συνεργασίας και είμαι βέβαιο ότι έτσι θα συνεχίσουμε, κυρία εισηγήτρια, με καλή θέληση και με λίγο παραπάνω χρόνο, νομίζω ότι θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε κάτι πολύ θετικό και ικανοποιητικό και για την εσωτερική αγορά και για τους συμπολίτες μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Λεγκρέιπ, ο κύριος Μπουζόη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι ο αριθμό των πολεμιών που κατατέθηκαν για αυτή την πρόταση οδηγία αποδεικνύουν τη σημασία της για τους επαγγελματίε και το ενδιαφέρον που προκαλεί. Θα στηρίξω λοιπόν την πρόταση της κυρίας Βερνιό να ψηφιστεί η πρόταση αυτή τον Ιανουάριο του 2013. Κάποιες πολύ σύντομες παρατηρήσεις. Θα προσπαθήσω να μιλήσω λιγότερο από πέντε λεπτά για το θέμα των συμβολιογράφων. Θα θυμάστε ότι έχω τοποθετηθεί για το θέμα αυτό επανειλημμένος. Απλώς θα περιοριστώ τώρα να πω ότι οι συμβολιογράφοι αναλαμβάνουν αρμοδιότητες από τις ε, δημόσιες αρχές που τις εκχωρούν. Δεν μου φαίνεται λογικό να μπορούν μια τέτοια εκχωρημένη αρμοδιότητα οι συμβολιογράφοι, ε, αρμοδιότητα εκχωρημένη από την Εθνική Αρχή ενός κράτους μέλους, να την εξασκούν και σε ένα άλλο κράτος μέλος. Δεν είναι οι υπηρεσίες τους της ίδιας φύσης με άλλες υπηρεσίες που κυκλοφορούν ελεύθερα εντός της νέας αγοράς. Θα έλεγα λοιπόν ότι πρέπει να αποκλειστούν πλήρω από το πεδίο εφαρμογή αυτή τη οδηγία. Για την ε, μερική πρόσβαση, νομίζω πρέπει να λάβουμε υπόψη τι προκλήσει ασφάλεια και προστασία των ε, ασθενών, οπότε θα πρέπει να μην ισχύουν οι διατάξει αυτέ για τα επαγγέλματα υγεία. Επίση, για τα επαγγέλματα του υγειονομικού κλάδου, θα πρέπει το σύστημα IMI να ισχύει εφόσον οι επαγγελματίε δεν έχουν πλέον το δικαίωμα να εξασκούν τα καθήκοντά τους μετά από τελεσίδικη απόφαση του αρμόδιου οργάνου προκειμένου να ε, γίνει συμβαστό και το τεκμήριο αθωότητα. Τώρα, για τι απαιτήσει, για τι ειδικεύσει, τι ιατρικέ ειδικεύσει, έχω καταθέσει τροπολογία που διευκρινίζει τι αρμοδιότητε που πρέπει να υπάρχουν και να αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια αυτή τη ε, περίοδου. Αυτό το έχει λάβει υπόψη η κυρία Βερνιό και για τι μέρε. Γιατί να μην κάνουμε το ίδιο και για του γιατρού και του οδοντιάτρου. Μιλάμε για τομείς όπου ε, απαιτούνται ειδικέ αρμοδιότητες όπως η πρόληψη, η εξέταση των ασθενών, η αγωγή που θα παρασχεθεί στον ασθενή και ούτω καθεξής. Θα πρέπει βεβαίως αυτά να τα ε, συζητήσει επισταμένως η Επιτροπή με τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες. Τώρα, για τις Πολωνές και Ουμάνες ε, νοσηλευτρίες, δεδομένου του κεκτημένου και των εξελίξεων στο εθνικό μας επίπεδο του πλαισίου κατάρτισης των νοσηλευτριών, δεν νομίζω ότι πρέπει να είναι δυσμενέ το πλαίσιο που ισχύει, δυσμενέ τώρα από το άρθρο 33. Για την κατάρτιση αυτή να σας δώσω κάποια στοιχεία πολύ σύντομα. Η αρχική εκπαίδευση στη Ρουμανία ήταν ήδη ιδιαίτερα ποιοτική, αλλά συμπληρώθηκε και από περαιτέρω διαβιωμάτιση. Από τα σχολικά ήδη χρόνια, από το 87-88 συγκεκριμένα, η αρχική ε, εκπαίδευση είναι τριετής, δηλαδή 4.600 ώρες. Πολλές ε, νοσηλεύτριες έχουν κάνει και εκπαίδευση μετά το σχολείο ε, και με συμπληρωματικά μαθήματα σε ειδικευμένα ιδρύματα. Αυτές οι νοσηλεύτριες πολλές φορές έχουν παρακολουθήσει και εκπαιδευτικά προγράμματα ε, για κάτι που αποτελεί υποχρέωση προκειμένου να εξασκούν τα καθήκοντά τους σε πολλές περιπτώσεις. Σύμφωνα με τις γνώσεις μου και τις πληροφορίες που μου δίνουν οι ρουμανικές αρχές ε, και υφυπουργό ε, στο Υπουργό Υγείας ε, στη Ρουμανία που βρίσκεται και στην αίθουσα μαζί μας, δεν γνωρίζει να υπάρχουν προβλήματα ιατρικών σφαλμάτων που να έχουν προκύψει από Ρουμάνες νοσηλεύτριες σε άλλα κράτη-μέλη. Οι νοσηλεύτριες αυτές που πρέπει να υποχρεώσουν να αποδείξουν την έχουν την υποχρέωση να αποδείξουν την επαγγελματική του πείρα για 5 συν 7 έτη, όπω και το άρθρο 33α τη οδηγία ορίζει, είναι 4.800 στον αριθμό. Δεν είναι μεγαλύτερο ο αριθμό. Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι θα πρέπει να εγγυηθούμε και στι νεσολεύτριε αυτέ την ίση μεταχείριση και να καταργηθούν οι επιπλέον απαιτήσει για την αναγνώριση των επαγγελματικών του προσόντων. Ιδάλω, οι νοσηλεύθερε αυτέ θα παραμείνουν σε μια κατάσταση δυσμενέστερη μέχρι να αναθεωρηθεί ξανά η οδηγία, κάτι που δεν ξέρουμε βεβαίως πότε θα συμβεί. Να ολοκληρώσω λέγοντας ότι για την ιατρική, καθώς και για τους επαγγελματίες, η εκπαίδευση δεν θα πρέπει να μετράται σε μονάδες ECTS. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα συμπληρωματικό εργαλείο, αλλά εφόσον δεν έχουμε μεμορφό σύστημα μέτρησης των μονάδων αυτών, θα πρέπει να είμαστε συναρτοί και προσεκτικοί. Θα πρέπει να δούμε κατά πρώτον την αναγνώριση των ακαδημαϊκών τίτλων. Τέλος, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την αρχική εκπαίδευση που έχει αποκτήσει κανείς το πρόγραμμα ενό κύκλου σπουδών ώστε να αποφύγουμε την επικάλυψη ισότιμων ε, προγραμμάτων σπουδών. Ακόμη και αν η συνέχεια του προγράμματος που ξεκίνησε σε ένα κάτω μέλος ολοκληρώθηκε σε ένα δεύτερο. Θα πρέπει να υπάρχουν ε, περιπτώσεις απαλλαγής. Αυτό ισχύει ως μηχανισμός για την ασυλεύτρια στο κείμενο. Θα πρέπει λοιπόν να επεκταθεί και σε άλλα επαγγέλματα του ιατρικού κλάδου κατά την άποψή μου. Σας ευχαριστώ κυρία Βερνιό. Ευχαριστώ και τους υπόλοιπους και όλους για την προθυμία τους και την επικοδομητική συζήτηση που είχαμε για να καταλήξουμε σε συμβαστικές λύσεις. Ελπίζω ότι θα έχουμε μια θετική ε, συμφωνία για να βελτιώσουμε την κινητικότητα των επαγγελματιών. Uh, thank you, Mrs. Ευχαριστούμε κύριε Μπουζόη. Κυρία Ρούλα. Ευχαριστώ πολύ. Σε πολλά σημεία συμφωνούμε γιατί όλοι θέλουμε περισσότερη και καλύτερη πρόσβαση, κινητικότητα, την ενίσχυση μιας ενιαίας αγοράς απασχόλησης. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το επιτύχουμε αν πάρουμε αποφάσεις που αντιτίθεται στα συμφέροντα των ίδιων των ενδιαφερομένων. Θα ήθελα να σας πω ότι όσον αφορά την εξέβρεση συμβαστικής λύσης, κάπου υπάρχουν κάποια όρια. Στη Γερμανία έχουμε συζητήσει με τους ειδικού του κλάδου, παραδείγματο χάρη ε, στον τομέα των νοσοκόμων, αλλά όχι μόνο των νοσοκόμων. Και η γενικότερη άποψη είναι ότι αυτή η αναθεώρηση της οδηγίας θα δημιουργήσει σε επιδείνωση της κατάστασης. Εάν λοιπόν δεν ε, συμμετάσχουν όλοι αυτοί οι ενδιαφερόμενοι σε αυτήν την προσπάθεια αλλαγής του κειμένου, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να πετύχουμε τίποτα. Και πολλές φορές βλέπουμε ότι από τη μία υπάρχουν πάρα πολλές δηλώσεις υπέρ αυτής της διτής εκπαίδευσης, του διτού συστήματος κατάρτισης. Από την άλλη, στην ουσία, όταν διαβάζει κανείς το κείμενο, διαπιστώνει ότι τίποτα τέτοιο δεν ακολουθείται στις αλλαγές του κειμένου. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να στείλουμε ένα μήνυμα θετικό όσον αφορά αυτήν την διτή κατεύθυνση στον τομέα της κατάρτισης, της εκπαίδευσης, γιατί είναι ένα πολύ ισχυρό μήνυμα όσον αφορά την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Θα πρέπει, επαναλαμβάνω, αυτή η μεταρρύθμιση να γίνει με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων. Θα πρέπει να είναι προαιρετική, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες να μπορέσουν να συμμετάσχουν, να κάνουν προτάσεις και να συμπεριληφθούν σε αυτή την αλλαγή. Αλλιώ, επαναλαμβάνω, αν δεν έχουν πρόσβαση στην προετοιμασία, δεν πρόκειται να πετύχουμε. Είναι πολλά τα θέματα που ακόμα πρέπει να συζητηθούν. Έρχομαι τώρα στο θέμα των νοσηλευτριών, παραδείγματος χάρη. Όλοι θέλουμε να αυξηθεί η ποιότητα. Όλοι θέλουμε να αναβαθμιστεί το σύστημα. Αυτό δεν είναι κάτι που μας χωρίζει. Αυτό που μας χωρίζει είναι ότι η αύξηση της διάρκειας της εκπαίδευσης είναι η πρόταση κάποιων. Κάποιον άλλον η πρόταση είναι να γίνει μια πιο ολοκληρωμένη αναβάθμιση και αναθεώρηση της κατάρτισής τους. Σχολικής, θεωρητικής αλλά και πρακτικής. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε λίγο πιο ευέλικτες λύσεις και κυρίως να συμμετάσχουν στην εξέβρεση λύσης και οι ενδιαφερόμενοι. Uh, thank you very much indeed. I just... Σας ευχαριστώ ειλικρινώς. Ο η κυρία Μακλάρκιν δεν είναι εδώ. Οπότε να επιμείνω στο σημείο που Δείξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον η ομάδα μου, συντηρητικοί και μεταρρυθμιστέ. Η κυρία Ρούλε μα είπε ότι η ευρεία εφαρμογή αυτή τη οδηγία σε σχέση με τα επαγγέλματα που θα είναι νομοθετικώ κατοχυρωμένα, και αυτό αφορά πολλά κράτη-μέλη, μπορεί να είναι δυσανάλογο και να δυσανάλογα να εμποδίζεται η πρόσβαση πολιτών άλλων χωρών. Διότι οι ανάλογε δομέ δεν λειτουργούν ανάλογα σε όλα τα κράτη-μέλη. Ε, αυτό το σχόλιο είναι πολύ καλή αφορμή για να πω ότι εμεί επιδιώκουμε τη βελτίωση τη κινητικότητα των επαγγελματιών και ώστε όλοι να μπορούν να εξασκούν τι δεξιότητέ του παντού. Η κυρία Μακλάρκιν έχει υποβάλει τροπολογίε για να επιταχυνθούν οι διαδικασίε και να μην υπάρχει η παρεμπόδιση εξάσκηση καθηκόντων από τα κράτη-μέλη βάσει τη εθνικότητα και τη ηθαγένεια. Ιδίω για σκοπού δημοσίου συμφέροντο συνθήκε εκπαίδευση. Όντω υπάρχουν διαφορέ μεταξύ των κρατών μελών, υπάρχουν διαφορέ μεταξύ των εκπαιδευτικών του συστημάτων και οπωσδήποτε το σύστημα θα πρέπει να επικεντρώνεται στο αποτέλεσμα, στο τελικό αποτέλεσμα και αυτό στην διαδικασία αυτή καθεαυτή. Αυτό αφορά τα περισσότερα επαγγέλματα και είναι ένα ζήτημα τη κατάρτιση γενικώ. Για τα επαγγέλματα του υγειονομικού κλάδου Νομίζω θα γνωρίζετε τι έχει ε, μελετήσει στην αρχική της έκθεση για, τις, ε, για τους γλωσσικούς ελέγχους και τους σχετικούς μηχανισμούς. Ε, νομίζω αυτό είναι σημαντικό για τους ασθενείς που μετακινούνται μεταξύ των κρατών μελών. Θα πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε τη δημόσια στήριξη και για την κινητικότητα των εργαζομένων, όμως αυτό μπορεί να υπονομευθεί από την πλημελή παρακολούθηση των επαγγελματικών προσόντων σε πολλές περιπτώσεις για την ε, κάρτα θα πρέπει να είναι νομίζω ένα εργαλείο οικειοθελούς χρήσης ε, το οποίο θα πρέπει να διατίθεται κατόπιν ετήσεως και να παράσχεται στους επαγγελματίες ώστε να βεβαιωθούμε ότι το κόστος θα είναι αναλογικό με την προσπάθεια. Επίση, οι αμοιβέ είναι κάτι που θα πρέπει να το καθορίζουν οι ενδιαφέρομένε αρμόδιε αρχέ. Κάτι που πάντοτε βέβαια θα πρέπει να διασφαλίζουμε όπω και στι άλλε περιπτώσει ότι θα είναι δυσανάλογο ω μέτρο και θα πρέπει να ακολουθήσουμε ρεαλιστική προσέγγιση. Μια συγκεκριμένη παρατήρηση που δεν αναφέρθηκε ακόμη. Έγιναν πολλά σχόλια για την εξέλιξη των επαγγελματικών κλάδων, ιδίω για το τι συμβαίνει με τι νοσηλεύτριε και γενικότερα στον ιατρικό κλάδο. Να θυμίσω ότι τον τομέα τη υγειονομικής περίθαλψη υπάρχει συνεχώ μεγαλύτερη πίεση για τι ειδικότητε. Ιδίω την ε, παρακολούθηση και την φροντίδα των ε, ηλικιωμένων. Εκεί πρέπει να υπάρχει καλή διοργάνωση των δεξιοτήτων που απαιτούνται από του επαγγελματίε και βεβαίω να διασφαλίζεται η προστασία των ασθενών. Κάτι που δεν συμβαίνει με τον ίδιο τρόπο σε όλε τι χώρε για τη μερική πρόσβαση. Νομίζω πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και εδώ η κυρία Μακλάκιν έχει υποβάλει τροπολογίε στην κατεύθυνση αυτών που πιστεύουν ότι εδώ πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Οι χειρισμοί μα πολύ επιλεκτικοί για την κατάρτιση της ε, ανανέωσης των επαγγελματικών ε, γνώσεων. Οι επαγγελματίες θα μπορούσαν με τον τρόπο αυτό να αποσβέσουν το κόστος της εκπαίδευσής τους αλλά το κόστος αυτός δεν θα πρέπει να είναι δυσανάλογο. Δηλαδή να μην χρησιμοποιείται ως ε, μέσο για να εμποδιστεί η είσοδος νέων επαγγελματιών στον κλάδο. Εδώ θα συνεχίσουμε να έχουμε εντατικές συζητήσεις με τα κράτη-μέλη για τη χρήση των κατεξουσιοδότηση πράξεων. Το επισημαίνει αυτό η κυρία Μακλάρκιν και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα απηχηθούν οι δικές μας υποθετήσεις και να υπάρχει απαραίτητος, ε, απαραίτητη διοργάνωση διαβουλεύσεων, η αναγκαία διοργάνωση διαβουλεύσεων προκειμένου να εγκρίνονται κάθε φορά για την εξοδότηση πράξη. Αυτό είναι το περιεχόμενο των τροπολογιών. Τώρα έχουμε πέντε λεπτά από τι προφορίε. Νομίζω μπορούμε να κλέψουμε λίγο χρόνο από τι προφορίε Είναι και πολλοί συνάδελφοι που θέλουν να παρέμβουν, αλλά θέλω να δώσω λόγο και στου κοιόδη. Mr. Kreutzmann, Mrs. Mrs. Now, can I ask you να σας παρακαλέσω να παραμείνετε στο δίλεπτο καθένας και η καθεμία σε αυτή τη φάση. Τη συζήτηση θα τη συνεχίσουμε και αργότερα, γιατί έχουμε ανταλλαγή απόψεων και στις 26 Νοεμβρίου. Οπότε θα μπορέσουμε τότε να δούμε τις συμβαστικές προτάσεις. Δύο λεπτά λοιπόν στον καθένα, το μέγιστο,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 θα μου επιτρέψετε δυόμιση λεπτά να χρησιμοποιήσω, γιατί είμαι εδώ από χθε, από την αρχή μέχρι το τέλο ε, τη συνέδρια. Λοιπόν, να πω κάποια πράγματα. Ε, αυτά που είπατε κι εσείς είναι αυτά που πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, πραγματικά να βλέπουμε πιο πολύ την έκβαση, το αποτέλεσμα, ιδίω στον τομέα τη υγεία και νομίζω ότι αυτό ισχύει και για όλου του ε, τομεί ε, της εκπαίδευσης κατάρτισης. Και αυτό που προτείνεται μέχρι στιγμή δεν εστιάζει εκεί. Όσον αφορά την δημιουργία διπλής πρόσβασης, διπλής δυνατότητας πρόσβασης, μπορεί να δημιουργήσουμε διακρίσεις. Εμείς κάναμε λοιπόν μια πρόταση συμβαστική που αποκλείει αυτή τη δυνατότητα διακρίσεων. Και οι δύο συνάδελφοι Ρούλε και Βάις προετοιμάσαν <clears throat> προετοιμάσαμε αυτήν την ε, πρόταση η οποία συμπεριλαμβάνει μία θεωρητική κατάρτιση, πανεπιστήμιο, το και την ίδια ώρα πρακτική. Σκοπός μας είναι η, ο αποκλισμός της κάθε δυνατότητας διάκρισης. Αντίθετα δηλαδή, όχι να δημιουργήσουμε διακρίσεις, αλλά να αποκλείσουμε τις διακρίσεις. Δεύτερον, αν κατάλαβα καλά τι είπατε, Μπορούμε να συζητήσουμε α, την πρότασή σας. Είπατε όσον αφορά τους συμβολιογράφους, θέλετε να δώσετε σε αυτό τον κλάδο τη δυνατότητα να παραμείνει στην χώρα από την οποία προέρχεται. Εδώ όμως αναφέρεστε στην ελευθερία παροχής υπηρεσιών, όχι εγκατάστασης. Δεν βοηθάμε λοιπόν τους συμβολιογράφους αν τους ε, αποκλείσουμε από την δυνατότητα να κινηθούν. Θα πρέπει να βρούμε μια εξαίρεση όσον αφορά την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, αλλά όχι εξαίρεση όσον αφορά την εγκατάσταση. Σε αυτή την περίπτωση θα υπόκεινται σε ένα εθνικό σύστημα. Αν κάποιος παντρευτεί με μία Πορτογάλ ή έναν Ισπανό, θα πρέπει να μπορεί να μην αποκλείεται λόγω της εθνικότητάς του. Και να μπορεί να υπόκειται σε όλες τις διατάξεις και τις προβλέψεις της χώρας στην οποία θα εγκατασταθεί. Επαναλαμβάνω λοιπόν, Όσον αφορά την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, ναι. Όσον αφορά την ελευθερία εγκατάσταση, εδώ θα πρέπει να μην του αποκλείσουμε. Συμφωνώ με αυτό που είπε η κυρία Ρούλε. Υπάρχουν σαφώ διαφορετικέ θέσει. Σε όλες τις χώρες αυτό δεν είναι απλώς εθνική η διαχωριστική γραμμή εδώ. Ευχαριστώ πολύ πάντως την εισηγήτρια γιατί έχει δείξει ανοιχτό πνεύμα και νομίζω ότι βρισκόμαστε σε καλή ε, οδό. Είμαι πολύ γενναιόδρο μαζί σα, ε, Ξεπεράστηκε και τα τρία λεπτά. Λοιπόν, κυρία Πέντρεγκαστ. Κύριε Πρόεδρε, θα ικανοποιηθείτε πολύ μαζί μου γιατί θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Και αυτό ήταν και το μισό που ήδη είπε. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω την Περναντέτ για την πάρα πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει και πιστεύω επειδή χθε ε, συναντήθηκα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Νησιλεπτών στην Κροατία, νομίζω ότι είναι σημαντικό να μην έχουμε αποδυνάμωση των διατάξεων για τις αρμοδιότητες και τα προσόντα των νοσηλευτεριών. Τα υπόλοιπα έχουν καλυφθεί. Ευχαριστώ. Um, uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε τα θέματα αυτά για να γνωρίζουμε ότι υπάρχει ενημέρωση διαρκώς μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι καταπληκτικό να έχουμε μια εισηγήτρια που τόσο καλά αντιλαμβάνεται το πόσο ζητιούνται τα θέματα αυτά και στην Επιτροπή που δείχνει ανοιχτή, ανοιχτό πνεύμα και που δημιουργεί ένα ισορροπό κείμενο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και για όλο μας την εργασία στην, ε, ε, και τις προσπάθειές μας στην Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, ήθελα να επικεντρωθούμε σε ό,τι επιτρέπει τη διευκόλυνση, την τόνωση, την ε, καλλιέργεια της κινητικότητας. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια αγορά δυνατοτήτων εργασίας στην Ευρώπη. Είναι ένα από τα σημαντικότερα καθήκοντα που έχουμε αναλάβει. Εδώ λοιπόν την επαγγελματική κάρτα, και εδώ ευχαριστώ την Κωνσταντς για τη στήριξή της, την βλέπω όχι ως έναν τρόπο να ρυθμίσουμε τους επαγγελματικού κλάδους, ούτε τα διοικητικά κόστη, τα, τους φραγμούς, αλλά έναν τρόπο να διευκολύνουμε την κινητικότητα. Σας παρακαλώ την τροπολογία μου 95, λοιπόν, συνάδελφοι, να την ε, υποστηρίξετε για το θέμα αυτό. Επίσης, να πω ότι η τροπολογία της κυρίας Μακλάρκιν που σχολίασε και ο κύριος ε, Χάρμπορ, είναι σημαντική. Υπήρξα σκιώδης ε, εισηγητρία για την έκθεση του κυρίου Μπίλαν για το σύστημα πληροφοριών. Είναι σημαντικό να αδράξουμε αυτή την ευκαιρία για να συμπεριληφθεί το θέμα και στην συγκεκριμένη περίπτωση. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε μου σύντομα γιατί είπαν πολλά ήδη οι συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κρότσμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε θα μιλήσω και εγώ για το θέμα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης. Όντως οι θέσεις εδώ από τη μία χώρα στην άλλη είναι διαφορετικές. Ξέρετε, οι Αμερικάνοι λένε ότι εδώ η ουσία είναι πιο σημαντική από την μορφή. Substance over form. Νομίζω ότι εδώ αυτό θα πρέπει να επικρατήσει και σε εμά. Άκουσα πολλούς από τους προηγούμενους ομιλητές. Ξέρω ότι πολλές φορές η Επιτροπή κάνει προτάσεις εμείς ε, στη Γερμανία έχουμε ένα σύστημα αρκετά ικανοποιητικό, αλλά βεβαίως θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί το σύστημα να λειτουργήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως είπε η κυρία Ρίλε, αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ να αναγνωρίζονται τα προσόντα, όποια και αυτά να είναι, στις άλλες χώρες. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να κάνουμε ένα περιοριστικό σύστημα, ένα σύστημα που θα αποκλείσει τους νέους και θα δημιουργήσει ακόμα περισσότερη ανεργία. Στον τομέα της υγείας, στον τομέα της νοσηλείας υπάρχει τεράστιο κενό, τεράστιες ελλείψεις και θα ήταν μεγάλο λάθος να περιορίσουμε την πρόσβαση των νέων σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σάλτεμοζε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ξεκινήσω ευχαριστώντα την εισηγήτρια για την εισηγήσή της. Ήταν ε, πολύ σημαντικό να, δούμε ένα, να βρούμε έναν τρόπο για να καλυφθούν όλες οι διαφορετικές απόψεις με συμβαστικές λύσεις. Υπάρχουν πολλοί που σχολιάζουν το διτό σύστημα, το τι μπορεί να συμβεί για τις με τις νοσηλεύτριε λόγω χάρη. Εδώ όμως δεν θέλουμε να διακυβευτεί το επίπεδο ή να αμφισβητηθεί το επίπεδο εκπαίδευση ή προσόντων των υπόλοιπων χωρών. Αν είναι πολύ ψηλό το επίπεδο για τι νοσοκόμε σε μια χώρα, θα πρέπει αυτό να ισχύει και για του υπόλοιπου. Θα πρέπει λοιπόν να, ε, γίνουν, ε, να γίνει αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων χωρί να αποδυναμώνεται ε, η εκπαίδευση στι χώρε που ειδήθηκαν τον υψηλό επίπεδο. Κυρία Βάιλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω στον κύριο Κρόιτσμαν, γιατί άκουσα προσεκτικά αυτά που είπε, εγώ ξέρω από δική μου εμπειρία πόσο σημαντικό είναι να αναγνωρίζει κανείς τα συστήματα και των άλλων. Το θέμα όμως εδώ είναι ότι κάποια πτυχία, κάποιοι τίτλοι που υπάρχουν, δεν μπορούμε να τους αμφισβητήσουμε ούτε να τους αγνοήσουμε. Εμάς μας ενδιαφέρει βεβαίως τα χρήματα που επενδύονται στους νέους στην κατάρτισή τους και στην εκπαίδευσή τους να οδηγούν σε μια καλή κατάρτιση. Στη Γερμανία έχουμε ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε εδώ να υποβαθμίσουμε τα επίσημα πτυχία και τίτλους. Στη Γερμανία, αν η πρόταση αυτή εφαρμοστεί, σίγουρα θα δημιουργηθούν μεγάλες αλλαγές. Υπάρχουν όμως και κάποιοι φορείς, κάποιες ενώσεις ενδιαφερομένων επαγγελματιών, οι οποίοι υποστηρίζουν αυτές τις αλλαγές. Αν λοιπόν βρούμε μια συμβιβαστική λύση, παραδείγματο χάρη 10 χρόνια συν 2 συν 3 και αυτά τα 2 ή 3 χρόνια επιπλέον κατάρτιση είναι ουσιαστική κατάρτιση, ε, σίγουρα αυτό θα μπορέσουμε να το υποστηρίξουμε. Σε καμία περίπτωση όμως δεν πρέπει από την πίσω πόρτα να ε, μπει ένα σύστημα το οποίο θα υποβαθμίζει την κατάρτιση που έχουμε πετύχει τόσα χρόνια στη Γερμανία με την πρακτική, με την πρακτική κατάρτιση συν την θεωρητική. Με 7 ή 8 χρόνια, εάν υποβαθμιστεί το σύστημα με έναν τρόπο πλάγιο, αυτό θα είναι πραγματικά πάρα πολύ αρνητικό για όλους μας. Κυρία Δαραμπέλα, θέλετε το λόγο γιατί καθυστερήσατε. Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Και εγώ είμαι υπερασπιστή ε, ε, του ανώτερου επίπεδου εκπαιδευτικών συστημάτων και έχω ασχοληθεί και με την ε, εκπαίδευση των νέων στο ανάλογο Βελγικό Υπουργείο. Ε, πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη όλες τις διαστάσεις της κατάρτισης, τι γίνεται με τις επιχειρήσεις και την ε, άσκηση εκεί, ε, πώς δυσκολεύεται κανείς να περάσει στον επαγγελματικό κόσμο και να ενταχθεί σε μία ομάδα. Πριν από δύο χρόνια λοιπόν ε, οργανώσαμε ένα διαγωνισμό για τα τεχνικά επαγγέλματα στο Βέλγιο το Βέλγιο δεν είχε τα καλύτερα αποτελέσματα. Οι χώρε που διακρίθηκαν περισσότερο ήταν η Γερμανία, η Αυστρία και η Φινλανδία και λιγότερο η Ελβετία. Που ε, είναι χώρε που καλλιεργούν την ε, εκπαίδευση τόσο στο ακαδημαϊκό επίπεδο όσο και σε ένα ε, επιχειρησιακό κλάδο. Ήμουν πολύ σύντομο λοιπόν, όπω θα τα σεβάστηκα την πίεση του χρόνου που έχουμε. thank Και σα ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί μα δώσετε και πολύ χρήσιμε πρακτικέ πληροφορίε. Γιώργεν Τίτσε, δυστυχώ ε, έχει πολύ λίγο χρόνο τώρα. Μπορεί να επανέλθει. Αλλά αν έχει ε, για δύο λεπτά κάποια σύντομα σχόλια, θα σου δώσω το λόγο και μετά θα δώσω το λόγο στην κυρία Βενιού για να κλείσουμε. Κύριε Στίτσερ, ευχαριστώ πολύ. Πολύ ευγενικό εκ μέρου σα που μα δίνετε και μα δύο λεπτά για να κάνουμε μια πρώτη εκτίμηση ε, των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί. Πρώτα απ' όλα, χαιρετίζουμε την υποστήριξη που δείχνει η Επιτροπή σα στην όλη αυτή η πρωτοβουλία και να μην ξεχνάμε ότι θα ήταν καλό για την ενή αγορά να ολοκληρώσουμε ε, στη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική περίοδο ε, το θέμα αυτό. Σε ό,τι αφορά τώρα την επαγγελματική κάρτα, να ξεκινήσω από αυτό, ήταν έτοιμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εμείς το ακολουθήσαμε πολύ μεγάλο ενθουσιασμό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θα πρέπει να δούμε τελικά, λαμβάνοντα υπόψη και τι ε, τροπολογίε που έχουν κατατεθεί, μπορούμε να προχωρήσουμε προ μια Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Κάρτα. Ναι, όταν έχει πραγματικά ως ε, αποτέλεσμα την απλούστευση. Και το θέμα της αναγνώρισης είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θα θέλαμε να παραμείνει αυτό το ε, σχήμα της σιωπηρής αναγνώρισης. Είναι θεμελιώδες και αυτό το μήνυμα θέλω να το μεταφέρω ξεκάθαρα προς εσάς. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα για τη μερική πρόσβαση. Θα ακούσουμε ε, πολύ προσεκτικά τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο για να δούμε αυτό το θέμα του αγκαντρεμό, καντράς της πλαισίωσης. Καλό θα ήταν επίσης ε, να κάνουμε και τη διάκριση μεταξύ των ε, house professionals και των professionals που δουλεύουν σε σχέση με το λεγόμενο security, ασφάλεια. Η τροπολογία 575 με ε, εξέπληξε κάπως. Είπαν και κάποιοι προλαλήσαντες κάποια σχόλια. Εμείς θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές σε ό,τι αφορά τις νοσηλεύτερες που βλέπω ότι εξαιρούνται με αυτή τροπολογία. Πρέπει να βρούμε πάντως ένα συμβεβασμό και για αυτό το σύστημα της διπλής εκπαίδευσης, διτής εκπαίδευσης. και για, κοινό, και για το κοινό πλαίσιο κατάρτιση. Πρέπει να προστατεύεται και αυτό θέλουμε και εμείς, θέλουμε να το προωθήσουμε. about... Να πω κάτι ακόμη για τις νοσηλεύτριες. Κατά την άποψή μας πρέπει να βρούμε συμβιβασμό. Ο Επίτροπος Μπαρνιέ είπε ότι θέλει να βρει μια, πραγματι... μια ρεαλιστική λύση, η οποία κατά την άποψή μας θα πρέπει να συνίσταται σε δύο στοιχεία. Πρώτον, ένα πολύ αυστηρό κατάλογο αρμοδιοτή, μάλλον ικανοτήτων και προσόντων ε, προσανατολισμένων στο αποτέλεσμα, αλλά να συμφωνήσουμε για τη διάρκεια. Αλλά σίγουρα να έχουμε αυτόν τον κατάλογο των προσόντων. Με εξέπληξε που για τις, για τις ε, ΜΕΕΣ δεν μίλησε κανένας. Κανένας δεν το ανέφερε αυτό για τη δωδεκαετία. Θέλω να το θέσω. Σε ό,τι αφορά τους γιατρούς, Έχουμε τροπολογίες, αλλά θέλω να σας ε, πω το εξής από αυτού. Στο τέλος, δεν θέλουμε να οδηγήσουμε σε ένα συμβιβασμό που θα σημαίνει όμως status quo, δηλαδή την οδηγία όσο έχει αυτή τη στιγμή, γιατί η οδηγία αυτή μέχρι στιγμής για τη βασική εκπαίδευση των γιατρών ε, προβλέπει διατάξεις πολύ δύσκολα μπορούν να εφαρμοστούν. Για τους συμβολογράφους την κυρία Βενιό και άλλους βουλευτές είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε για να καταλήξουμε σε συμβιβασμό, διότι δεν βλέπουμε ότι θα υπάρξει μεγάλη πρόοδο σε αυτό το θέμα. Πρέπει να υπογραμμίσω και ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Μπουσό. Για τους δικαστές δεν μπορούμε να έχουμε τους πελάτες να πληρώνουν τους δικαστές, αν θέλετε να το πω έτσι. Και υπάρχουν και κάποια κράτη που διατηρούν κάποιε απαιτήσει περιθαγένεια. Ίσως χρειαστεί να λάβουμε και περαιτέρω νομική δράση ως Επιτροπή. Μήπως μια ρήτρα αναθεώρησης ή ε, ε, μια ρήτρα αναμονής, ε, standstill clause, θα ήταν η λύση. Θα το δω με, το, με την ισχύτρια και του Σκιώδης, μήπως βρούμε μια λύση. Τέλος, ένα θέμα που επίσης δεν αναφέρθηκε. Βλέπουμε ότι υπάρχουν τροπολογίες που περιορίζουν σημαντικά την προσωρινή κινητικότητα. Τροπολογίες που έχουν κατατεθεί από και τους βουλευτές. Αυτό το καθεστώς προσωρινής ε, κινητικότητας είναι ένα νέο καθεστώς το οποίο εισήχθη από την το 2005 και νομίζω ότι είναι ένα στοιχείο που θα μας δώσει ανάπτυξη. Συμβάλλει στην ανάπτυξη αυτό το προσωρινό καθεστώς κινητικότητας. Δεν θέλουμε λοιπόν να πάμε προς τα πίσω. Σίγουρα θέλουμε να έχουμε έναν έλεγχο των προσόντων, παραδείγματος χάρη, ε, για τους ξεναγούς, κάποια πράγματα τα οποία προτείνονται. Όλα αυτά πηγαίνουν ε, αντίθετα από το στόχο μας που είναι η μεγαλύτερη ανάπτυξη. Πάντως θα προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε με την εισηγήτρια για να βρούμε λύσεις στα προβλήματα και θέλω να σας ευχαριστήσω που μου δώσετε το λόγο. Uh, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ γιατί πάντοτε είστε πάρα πολύ ξεκάθαρος σε αυτά που μας λέτε. Είστε και πάρα πολύ ντόμπρο και μας βοηθάτε με αυτό. Λοιπόν, κυρία Βερνιό έχει τώρα το λόγο πάρα πολύ σύντομα για να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Να ευχαριστήσω όλους τους αδέλφους που έλαβαν σήμερα το λόγο. Πραγματικά θα ήθελα να πω ότι η επιθυμία μας να βελτιώσουμε να δώσουμε περισσότερες δυνατότητες ε, στους Ευρωπαίους πολίτες αλλά και στους επαγγελματίες των κλάδων αυτών είναι κάτι που είναι πραγματικά μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρόκληση. Ελπίζω να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε αυτό το καλό κλίμα προς το γενικό συμφέρον όλων. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτώ το χρονοδιάγραμμα, βέβαια τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν και μπορούμε να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Επειδή ακόμα η αίθουσα είναι γεμάτη, παρακαλώ πολύ, ακούστε με. Αν θέλετε να φύγετε, μπορείτε να φύγετε με ησυχία, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Και θέλω να ευχαριστώ την κυρία Βάιλερ. Κυρία Βάιλερ, με ακούτε? Ήθελα να σας ευχαριστήσω που προεδρεύσατε χτες. Έμαθα ότι το κάνατε με εξαιρετικά κομψό τρόπο. Και επίσης ε, όσον αφορά την ακρόαση στην οποία θα πρέπει να εκπροσωπηθεί, στην οποία εκπροσωπήθηκε η Επιτροπή μας για θέματα εσωτερικής αγοράς που οργάνουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την Αρμόδια Επιτροπή, θα ήθελα να ξεκινήσουμε καταρχήν όσον αφορά την συνάρτηση που θα γίνει από τις 3 ως τις 6 την επόμενη εβδομάδα, την Τρίτη, θα προεδρεύσω επίσης τη συνάντηση αυτής. Νομίζω ότι οι πολιτικές ε, ομάδες γνωρίζουν τι διευθετήσεις έχουν γίνει για τη συνάντηση αυτή. Ο υποψήφιος επίτροπος ε, είναι τον Ιμπόγκ είναι σήμερα εδώ στις 11.30 θα εγκαταλείψω την ε, συνεδρίαση για να τον συναντήσω. Επίσης έχουμε ένα νέο μέλος ε, που προέρχεται από τη Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΤ. Την ε, καλωσορίζουμε εδώ και ελπίζω θα μας βοηθήσει και θα μας εμπλουτίσει με πολλά στοιχεία και μυστικά από τη Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΤ. Προχωρούμε λοιπόν στις ε, ψηφοφορίες. Το πρώτο θέμα είναι οι τιμές των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση. Ο εισηγητής είναι παρόν, έχετε όλες τις κάρτες σας. Υπάρχει εδώ κάποιος επικεφαλής, η Μπερναντέτ, για τους σοσιαλιστές, για τις ψηφοφορίες. Αλλιώς θα το κάνω εγώ. Συγγνώμη, δεν σας άκουγα, Πρόεδρε εσύ κατευθύνεις την ε, ψηφοφορία. Ναι. Δεν ξέρω, να ξέρω ποιον κοιτάω. 39. Υπέρ. Τροπολογία 39. Υπέρ. Κατά. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε την 39 αρχή της ψηφοφορίας για να ελέγξουμε. Λοιπόν, κυρία Βάιλερ, υπέρ, Τιμ κατά. Ωραία, εντάξει θα προσαρμόσουμε. 40 Χατζημαρκάκης. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 41 Φόξ. Υπέρ. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Τέλος. Εγκρίνεται. 42, Fox, αρχή της ψηφοφορίας. Τροπολογία 42. Τέλος. Εγκρίνεται. 43 καταπίτη. 44 βερνιό. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 5 συγητής. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 45 Βερνιό υπέρ. Α, ψηφίζουμε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τη 45. Τέλος, απορρίπτεται. 6 Μπεζόη υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 7 εισηγήτης υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 46 και 47 είναι ταυτόσημες, υπέρ, κατά, εγκρίνονται. 48 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 49 βερνιό. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 49. Τέλος. Απορρίπτεται. 8 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 50 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 51 βερνιό υπέρ. Ψηφίζουμε την 51. Τέλος. Απορρίπτεται. 52 της κυρίας Βερνιό. Ψηφίζουμε την 52. Τέλος. Απορρίπτεται και αυτή. 53 έχει αποσυρθεί. Ναι. 54 της κυρίας Βερνιό ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. 9. Του εισηγητή υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 55. Βερνιό. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τέλος. Απορρίπτεται. 56 Βερνιό. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Απορρίπτεται με δύο ψήφους διαφορά. 57. 57 της κυρίας Βερνιό. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Απορρίπτεται και αυτή. 10 του εισηγητή υπέρ. Κατά εγκρίνεται 58 βερνιό. Ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται 59 της κυρίας Βερνιό. Ψηφίζουμε. Τέλος. Και αυτή απορρίπτεται. 11 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 60 υπέρ κατά εγκρίνεται 61 ψηφίζουμε την 61 τέλος απορρίπτεται 12 του εισηγητή υπέρ κατά εγκρίνεται 62 Μπερνιό ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τέλος απορρίπτεται 13 του εισηγητή υπέρ κατά εγκρίνεται. 63 Βερνιό. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τέλος. Απορρίπτεται. 64 Βερνιό. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Απορρίπτεται. 65 Βάισκεβερ. Υπέρ. Κατά. Έλεγχουμε. 65 αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίνεται. 66 Βερνιό. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Απορρίπτεται. 14 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 69 Βερνιό. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Μπορείτε να ψηφίσετε λίγο πιο γρήγορα. Τέλος. Απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά. Αν κάποιο δεν ψήφισε, θα μπορούσε να έχει ανατραπεί το αποτέλεσμα. 15 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Δύο ταυτόσημες, που είναι και προσθήκη. 67 και 68 υπέρ, κατά, εγκρίνονται. 6, συγγνώμη, 16, 16, του εισηγητή. Υπέρ κατά εγκρίνεται 70 και 71 υπέρ κατά εγκρίνονται 72 και 73 υπέρ κατά εγκρίνονται 74 έχει αποσυρθεί 75 υπέρ κατά εγκρίνεται 76 έχει αποσυρθεί 77 Επίσης 17 του εισηγητή υπέρ. Κατά. συγγνώμη, υπέρ, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 78 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 79 υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. 80-81 καταπίπτουν γιατί εγκρίθηκε 17, 82 υπέρ, κατά, εγκρίνεται, 83 υπέρ, κατά, εγκρίνεται, 84 βερνιό υπέρ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 84. Τέλος. Απορρίπτεται. 85. Ψηφίζουμε την 85. Τέλος. Απορρίπτεται. 86. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 87. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 88. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 18 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται 89, Βερνιό. Ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. 90 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 91 Βερνιό. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Απορρίπτεται. 90 95 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 92 έως 96 καταπίπτουν. Η επόμενη έχει αποσυρθεί. 19, 98. Επίσης 99 υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Οι άλλες καταπίπτουν. 102. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 102. Τέλος. Απορρίπτεται. 103. 104. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 103 και την 104. Απορρίπτεται. 106 υπέρ. Ελέγχουμε. Όχι. Κατά. Δεν είναι ξεκάθαρο το αποτέλεσμα. Ψηφίζουμε την 106. 106. Τέλος, εγκρίθηκε. 105 έχει αποσυρθεί, 20 καταπίπτει, 108 υπέρ, κατά. 108 108 υπέρ, υπέρ της 108. Κατά. Πρέπει να ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 108. Τέλος, εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. 109 έχει αποσυρθεί, 110. 110 Υπέρ. Υπέρ της 110. Κατά. Απορρίπτεται. 111 έχει αποσυρθεί. 21 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 112. Ψηφίζουμε την 112. Τέλος. Απορρίπτεται. 113. 113 ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. 115 υπέρ. Ψηφίζουμε την 115 αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Απορρίπτεται η 115 με μικρή διαφορά. 22 του εισηγητή υπέρ. Υπέρ. 22. Είστε υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 114. Καλπέρτς. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τέλος, εγκρίθηκε με μία ψήφο διαφορά. 116. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ω, συγγνώμη, εγκρίνεται. 23 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 117 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 118 υπέρ κατά εγκρίνεται. 24 του εισηγητή υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 25 βερνιό υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 26 μπουζόι υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 27 βερνιό υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 28 γκρεκ υπέρ κατά εγκρίνεται. Η μία καταπίτη 30 χατζημαρκάκης υπέρ κατά απορρίπτεται. 29 φόξ υπέρ ελέγχουμε. Αρχή της ψηφοφορίας 29. Τέλος. Εγκρίνεται 29. 31. Αρχή της ψηφοφορίας, τροπολογία 31. Τέλος. Εγκρίνεται η 31. 2. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 3. Υπέρ. Κατά. Και αυτή εγκρίνεται. 35 έχει αποσυρθεί. 32. Φόξ. Υπέρ. Αρχή της ψηφοφορίας για την 32. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίνεται. Αυτό σημαίνει ότι οι άλλες δύο καταπίπτουν. Τέσσερα Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 36, 37 και 38. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται και οι τρεις. Ψηφίζουμε το σχέδιο γνωμοδότησης, το σύνολό του, με ηλεκτρονική ψηφοφορία, αρχή της ψηφοφορίας για το σύνολο του κειμένου, τέλος, 37 υπέρ, καμία ψήφος κατά. Ευχαριστούμε πολύ τον εισηγητή. Συγχαρητήρια. Και θα σταλεί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Περνάμε τώρα στην έκθεση της κυρίας συγγνώμη ο συνάδελφος ο κύριος Γκαρθές Ράμος πρόεδρε να αναγγείλω την απόσταση των τροπολογιών 53-54 και 50 Ωραία. Το λαμβάνουμε υπόψη, το καταγράφουμε. Να σας θυμίσω ότι εδώ συνεχίζεται το ηρωικό έργο εκ μέρους της Επιτροπής μας, της κυρίας Ρόιτοβα, που ασχολείται με την αναρμόνιση μια σειρά νομοθεσιών. Και περιμέναμε στο Συμβούλιο να υπάρξει γνωμοδότηση. Ε, Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων επίση έχει επιβεβαιώσει τη θέση τη για την επαναδιατύπωση αυτών των οδηγιών. Ε, η συγκίτρια θέλει να πει κάτι πριν ε, αρχίσουμε την ψηφοφορία. Κύριε Ρότοβα. Θα ζητήσω να τον λόγο μετά την ψηφοφορία, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ε, Ωραία, λοιπόν. Να περάσουμε στην οδηγία για τα όργανα μέτρησης κατά πρώτον. Να δούμε μερικές από αυτές τις τροπολογίες σε ομάδες. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν. Περνάμε ακριβώς στο, στην οδηγία για τα όργανα μέτρησης. 27, 29, 30, 31, 32. Θα τις ψηφίσουμε όλες μαζί. Συμφωνείτε. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. 33 της κυρίας Βερνιό. Άρχεται η ψηφοφορία για την 33. Πέρας. Μπορούμε να επιταχύνουμε. Απορρίπτεται. 8 της κυρίας Ρόιτοβα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35 της κυρίας Βερνιό. 25 της κυρίας Βερνιό. Εγκρίνεται. Ε, άρχεται ψηφορία. Can you please speed up your voting, because we are a bit short of time. All you need to do is press the button for me. Μπορείτε να επιταχύνετε λίγο Ωραία λοιπόν, απορρίπτεται. Άλλη ομάδα τώρα. 36, 37, 38, 39 και 41 μαζί. Υπέρ. Είστε κατά. Όχι, ωραία, όλες μαζί. Ομάδα δροπολογιών. Άρχεται η ψηφοφορία. 36, 37, 38, 39 και 41. Πέρας εγκρίνονται. 42 της κυρίας Βερνιό. Άρχεται η ψηφοφορία για τα 32. 42, συγγνώμη. Πέρας. Απορρίπτεται. Οι υπόλοιπε τροπολογίες που δεν έχουν αποσυρθεί. Δηλαδή 43, 50, 50 και 57 Εντάξει. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Και τέλος ψηφίζουμε το σχέδιο πρότασης, το σχέδιο ψηφίσματος. Στην τελική του μορφή άρχεται η ψηφορία. Παρακαλώ ψηφίστε. 37 κάρτες βλέπω. Κάποιος λείπει και δεν έχει ψηφίσει. Πέρας. 36 υπέρ, κανείς κατά. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα. Ο κύριος ε, Ραμόν έχει αποσύρει τις τροπολογίες του. Οπότε ψηφίζουμε την τροπολογία 35 της κυρίας Άλτε Μόζε. vote Πέρας. Απορρίπτεται. Η 54 αποσύρεται. Και τώρα μαζί η 9, 12, 10, 11, 13 μαζί. Εντάξει, καλά, όχι μαζί. 9 και 12 από κοινού. Υπέρ. Κατά. Άρχεται η ψηφοφορία. 9 και 12 μαζί. Uh, the vote is closed. Πέρας εγκρίνονται. 10. Υπέρ. Να δούμε αν μπορούμε να πάμε πιο γρήγορα. 10. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται με διαφορά. 11. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 13. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 14. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 56. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται με διαφορά. 16. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 57 ως προστίκη. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 17. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 18 και 19. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. 20. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 21. Ως προσθήκη. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 26 το αντίστοιχο τμήμα υπέρ κατά εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά εγκρίνεται. 33 να τις δούμε αυτές ε, από κοινού. 33. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 35. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 39. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 43. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά εγκρίνεται 67-69 αποσύρονται όχι την 69 δεν ψηφίσαμε υπέρ κατά εγκρίνεται 46 υπέρ κατά εγκρίνεται 47 ε, τεχνική τροπολογία 70 αποσύρεται ε, για τις ατολικές σκέψεις 1 υπέρ κατά εγκρίνεται 49 υπέρ κατά εγκρίνεται η 50 αποσύρθηκε 51 υπέρ κατά εγκρίνεται 3 υπέρ κατά επίσης εγκρίθηκε περνάμε στην τελική ψηφοφορία Άρχεται η ψηφοφορία. Άλλος κανείς, πέρας. Εγκρίνεται με 35 ψήφους υπέρ, καμία ψήφους αρνητική. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ρόιτοβα, θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για να ολοκληρωθεί η ψηφοφορία. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που με βοήθησαν για την επεξεργασία αυτής της δέσμης αναθεώρησης, καθώς και τη γραμματεία της ΣΥΜΚΟ και τους ε, βοηθού που μου επέτρεψαν να συνέβαλα μάλλον στην άσκηση πίεσης προς το Συμβούλιο. Ήταν χωρίς προηγούμενο η κατάσταση που δημιουργήθηκε. Το Συμβούλιο μας ε, μπλόκαρε για ένα εξάμεινο. Διότι δεν γνωμοδοτούσε. Επί έξι μήνε δεν είχαμε τοποθέτηση από το Συμβούλιο μέσω τη επιτοπολογία επί της έκθεσης μας. Έλεγαν ότι όλα πάνε καλά. Θέλω λοιπόν να ζητήσω εντολή από την Επιτροπή μας για να μπορέσω να την με την Κυπριακή Προεδρία για την επόμενη φάση της ανάγνωσης και να επιτύχουμε συμφωνία. Ελπίζω ότι θα μπορέσει η νομοθεσία αυτή να εγκριθεί ως τα Χριστούγεννα, εάν μου δώσετε εντολή. Δεν ξέρω αν με ακούγατε, Πρόεδρε, διότι ζητώ εντολή, εντολή για να αρχίσουν οι διαπραγματεύσει με την ε, Προεδρία. Διότι το πακέτο αυτό για τα αγαθά για το 2008 θα πρέπει να αρχίσει να φτάνει και στις επιχειρήσεις. Πρόεδρος, οι ε, συντονιστές συζήτησαν ε, την, το έτοιμά σας για εντολή και συμφώνησαν. Περιμένα να δούμε τι θα γίνει με την ψηφοφορία. Ελπίζω λοιπόν ότι ήλπιζα ότι θα το είχατε πει ευθύ εξ αρχή. Θα το είχατε θέσει το ζήτημα, γιατί ήθελε να είναι όλοι εδώ. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν τα μέλη τη Επιτροπή αν είσαστε υπέρ τη εντολή αυτή. Η κυρία Σαλντεμόζα, από ό,τι βλέπω, είναι παρούσα και είναι υπέρ. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικώ για την εντολή τη κυρία Ρόιτοβα. Πόσου χρειαζόμαστε, 21. Δεν είναι όμω όλοι εδώ τώρα. Λυπούμε, αλλά Έπρεπε να το έχετε θέσει πριν την ψηφοφορία. Δεν είναι αρκετή εδώ. Μπορούμε να βρούμε άλλου τρει για να ψηφίσουν. Πόσου χρειαζόμαστε, 21. Μπορείτε να βρείτε κάποιον να έρθει να ψηφίσει γρήγορα. Μπορείτε να βουτήξετε κάποιον απ' έξω να έρθει μέσα. One person. Everyone... Ένας φτάνει. How many people do we 40, 40 if you want. I need your vote. Yeah, okay. Just, that's all right. Okay, that's good. Somebody, somebody who's got the card in has not voted. Bernadette, can you just... Κάποιος έχει την κάρτα του στο μηχάνημα αλλά δεν έχει ψηφίσει. δεν μπορεί να ψηφίσεις. Ωραία. Λοιπόν, έχετε την εντολή σας, κυρία Ρωτόβα. Τη πήραμε τις 21 ψήφου. Μπράβο σα. So, Οι μελλοντικοί συγκεκριτές να είναι βέβαιοι ότι υπάρχουν αρκετοί στην αίθουσα. Σα ευχαριστώ πολύ λοιπόν όλους. Θα δούμε διαφάνειες τώρα, σωστά. Μισό λεπτό να ετοιμαστεί η παρουσίαση. Και είναι και ο κύριος Κομφεράτη, ο κύριος Μάντερς, που δεν ξέρω θα μιλήσει εκ μέρους των Πρασίνων. Ε, έχω κάποιες παρατηρήσεις από την κυρία Μακλάρκιν, ο κύριος ε, Γκυγιόν έχει φύγει. Θα ακούσουμε κάποια σχόλια για το θέμα αυτό και επίσης ελπίζουμε να έχουμε έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής. Uh, I should, uh, Μα συγχωρείτε που δεν καλωσορίσαμε την κυρία, την εκπρόσωπο τη Κυπριακή Προεδρία. Παρακολουθεί την εξέλιξη τη δέσμη μέτρων με πολύ προσοχή. Σα ευχαριστούμε λοιπόν που είστε εδώ. Ο κύριο Φαμπ θα μα κάνει την παρουσίαση. Εγώ θα πρέπει να αφήσω την Προεδρία, γιατί έχω συνάντηση, αλλά το όλο θέμα το παρακολουθώ και εγώ πολύ στενά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για μια έκθεση πρωτοβουλία. Θα σας παρουσιάσω σήμερα το σχέδιο όσον αφορά το θέμα της διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς. Πολλές συζητήσεις έχουν ήδη γίνει, επικοδομητικές, με τους κοιόδους συζητητές, καθώς και με τους εκπροσώπους ε, των ε, πολιτικών ομάδων. Ε, θα ήθελα να σας κάνω μια σύντομη παρουσίαση του πώς έχουν τα πράγματα σήμερα. Ευχαριστώ την κυρία Ποζίτσα την, από τη Γραμματεία, η οποία πραγματικά με στήριξε, καθώς και την συνεργάτη μου, την κυρία Μπέγκμαρ. Όσον αφορά τις ρυθμίσεις και τους κανόνες που υπάρχουν, στην Ευρώπη και ισχύουν σήμερα προβλέπουν ότι βεβαίως υπάρχει ίση μεταχείριση μεταξύ των ε, κρατών μελών. Διαπιστώνουμε όμως όλο και περισσότερο ότι πολλές φορές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξέρει, όχι πάντα όμως, ότι σε όλες τις χώρες, σε όλα τα κράτη-μέλη υπάρχουν οδηγίες οι οποίες δεν υλοποιούνται, δεν εφαρμόζονται σε κάποια κράτη-μέλη. Είτε εφαρμόζονται μερικώς. Θα ήθελα να σας πω καταρχήν ότι προσπάθησα να βρω μοντέλα μέτρησης, στοιχεία οικονομικά, τα οποία να μας δίνουν αποτελέσματα όσον αφορά την ενιαία αγορά και το κατά πόσον αυτή η ενιαία αγορά οδήγησε σε μια ανάπτυξη, σε πραγματικά αποτελέσματα. Και πραγματικά διαπίστωσα ότι αυτά τα αποτελέσματα δεν υπάρχουν. 0,8% περισσότερη ανάπτυξη. Αυτό είναι, αν θέλετε, το αποτέλεσμα που διαθέτουμε με πολλές βεβαίως δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης και βελτίωσης αυτών των αποτελεσμάτων. Εγώ καταρχήν λοιπόν σαν γενική διατύπωση θα ήθελα να πω, διαπίστωση, θα ήθελα να πω ότι μας ενδιαφέρει να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να έχουμε απτά αποτελέσματα, μετρήσιμα αποτελέσματα για την προστιθέμενη αξία αυτής της ενιαίας αγοράς. Και αυτό βεβαίως γιατί με δημοκρατικό τρόπο θέλουμε να παίρνουμε κάποιες αποφάσεις οι οποίες να εφαρμόζονται με ενιαίο τρόπο σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Υπάρχουν εδώ λοιπόν πολλές προτάσεις για το πώς μπορεί να γίνει καλύτερη ε, ενιαία εφαρμογή αυτών των δημοκρατικών αποφάσεων και γι' αυτό και αυτό που τελικά θέλουμε να εντοπίσουμε τα στοιχεία αυτά τα οποία είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει καλύτερα η ενιαία αγορά. Γι' αυτό και έχω λοιπόν κάνει κάποιες προτάσεις έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια καλύτερη διακυβέρνηση, καλύτερα αποτελέσματα, καλύτερη υλοποίηση, εφαρμογή, έτσι ώστε να υπάρξει καλύτερη μεταφορά των ε, ευρωπαϊκών, των κοινοτικών ε, νομοθετικών κειμένων, οδηγιών και άλλων σε εθνικό επίπεδο, με ενιαίο τρόπο με καλύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ έχει πολύ περιορισμένες δυνατότητες καθότι μπορεί να διαπιστώσει κάποιες ε, παραβάσεις στη συνθήκη και να ξεκινήσει μια διαδικασία επί Μπορούμε λοιπόν ήδη να στηριχτούμε σε αυτή τη δυνατότητα που έχει η Επιτροπή, αλλά μας ενδιαφέρει καταρχήν να υπάρξει περισσότερη διαφάνεια. Ένας επιπλέον στόχος που έχω εντοπίσει και έχω διατυπώσει είναι τα κράτη-μέλη τα οποία συμμετέχουν στη δημοκρατική διαδικασία απόφασης στο τέλος της αλυσίδας να εφαρμόσουν αυτά τα οποία έχουν αποφασίσει. Μήπως μπορείτε να βάλετε στην οθόνη την επόμενη διαφάνεια. Σας ευχαριστώ. Όχι αυτή, την επόμενη. Εδώ, αυτή, μάλιστα. Εδώ λοιπόν είναι πολύ σαφές αυτό που εγώ προτείνω. Πρώτον, περισσότερη διαφάνεια όσον αφορά την σημερινή κατάσταση. Πώς έχει η κατάσταση όσον αφορά τη μεταφορά των ευρωπαϊκών νομοθετικών κειμένων. Χρειαζόμαστε επίσης περισσότερες κατευθυντήριες γραμμές σε ευρωπαϊκό επίπεδο και βεβαίως από τη στιγμή που δεν υπάρχει ένα, αν θέλετε, κεντρικό σύστημα, να θέσουμε ενιαίους στόχους και κατά την άποψή μου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ καλείται να παίξει ένα ρόλο ελέγχου, συστηματικό έλεγχο όσον αφορά αυτά που έχουν ήδη αποφασιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν δηλαδή αυτές οι ήδη αποφασισμένες με δημοκρατικές διαδικασίες οδηγίες εφαρμόζονται πραγματικά στα κράτη-μέλη και από τα κράτη-μέλη. Έχουμε την εντύπωση σήμερα ότι είναι πιο εύκολο να ελέγξει κανείς την εφαρμογή νέων οδηγιών σε σχέση με τις πιο παλιές. Επίσης, θεωρώ ότι χρειάζεται περισσότερη ε, εποπτεία, επιτήρηση μεταξύ των κρατών μελών. Το ένα κράτος μέλος δηλαδή μπορεί να μάθει, να βοηθηθεί από το τι έκανε ένα άλλο κράτος μέλος. Κράτη-μέλη με περισσότερη εμπειρία μπορούν να βοηθήσουν νεότερα κράτη-μέλη. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμμετάσχουν τα εθνικά κοινοβούλια σε αυτήν τη διαδικασία εφαρμογής. Και σε πολύ πρώτα στάδια της διαδικασίας τα εθνικά κοινοβούλια να συμμετάσχουν και θεωρώ εδώ ότι η συμμετοχή τους θα βοηθήσει πάρα πολύ την περαιτέρω εφαρμογή αυτών των αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια καλύτερη οργάνωση αυτής της διαδικασίας Μιλήσαμε επί έναν πίνακα αξιολόγησης για τα αποτελέσματα της εθνικής αγοράς. Ένα σύστημα που ίσως να φέρεται περίπλοκο είναι όμως αν θέλετε ε, μία αξιολόγηση του τι έχει γίνει σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά την υλοποίηση αυτών των ε, αποφάσεων. Πίνακες αντιστοιχίας, αν θέλετε, οι οποίοι βεβαίως ε, την ίδια ώρα θα συμπληρώνονται και με κάποια στοιχεία που αφορούν την ανάπτυξη, την ετήσια ανάπτυξη στο κοινοβούλιο της κάθε χώρας πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες ημερομηνίες οι οποίες να συμπεριλαμβάνονται στο χρονοδιάγραμμα της κάθε προεδρίας που θα μετρώνται αυτά τα στοιχεία. Εμείς θα πρέπει να διασφαλίσουμε επίσης ποιες είναι οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την μακροοικονομική ανάλυση, και να μην αποκλειστεί εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από αυτή την παρακολούθηση ε, των στοιχείων αυτών και των στόχων αυτών. Κάποια στιγμή δηλαδή μεταξύ Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες συστάσεις για τις χώρες, country specific recommendations, που θα αφορούν την πρόθεση των στόχων που αφορούν την ενιαία αγορά αυτός ο πίνακας βαθμολογίας και οι πίνακες αντιστοιχίες όσον αφορά ε, τις επιδόσεις της ενιαίας αγοράς, αυτό είναι κάτι που εμάς εδώ στην, Ευρωπαϊκή, ε, στην ε, Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ενιαία Αγορά μας έχει αποσχολήσει εδώ και χρόνια. Πώς δηλαδή μπορούμε να μετρήσουμε την ε, αποτελεσματικότητα αυτών των αποφάσεων, πώς μπορούμε να παρακολουθήσουμε την μεταφορά σε εθνικό επίπεδο όλων αυτών που τον αποφάσουν. Και εδώ ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σαν στην συναπόφαση έχει παίξει και μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο. Υπάρχουν, όπως ξέρετε, πολλοί οι οποίοι επιθυμούν αυτή η διαδικασία να γίνει πιο επίσημη και βεβαίως ε, να καταλήξει σε μια έκθεση πρωτοβουλίας. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ξέρετε, προετοιμάζει τις, και αποφασίζει, ψηφίζει, τις κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά την πρόοδο στην ενιαία αγορά. Και τελικά βλέπουμε ότι ο ρόλος εδώ της Επιτροπής είναι καθοριστικός. Ο ρόλος Βεβαίω του Συμβουλίου δεν θα πρέπει εδώ να υποτιμηθεί σε καμία περίπτωση όσον αφορά την νομοθεσία που αφορά την ενιαία αγορά. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ εγώ ότι αυτό το άρθρο 26.3 θα πρέπει να θεωρηθεί σαν μια ικανή, ε, ισχυρή βάση, στηριζόμενη όμως πάντοτε και στη νομική βάση της κάθε οδηγίας ή του κάθε κανονισμού, κάτι που φυσικά θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συμπεριλαμβάνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από νομικής απόψεως, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθεί υπόψη. Άρθρο 26.3 λοιπόν, σε συνδυασμό πάντα με τη νομική βάση της κάθε οδηγίας, του κάθε κανονισμού, κάτι που θα ενισχύσει εδώ το ρόλο συναπόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όσον αφορά τη νομική βάση για ε, μια έκθεση πρωτοβουλίας νομοθετικού περιεχομένου, κάτι το οποίο θέλουμε να ε, συζητηθεί. Και ξέρω ότι αρχικά η διάσκεψη των Προέδρων αντέδρασε κάπως επιφυλακτικά. Πολλοί όμως ισχυρά επιχειρήματα ακούστηκαν και συζητήθηκαν και πιστεύω ότι εμείς σαν ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σίγουρα θα πρέπει να προωθήσουμε αυτή τη διαδικασία προς την ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συναπόφαση και σε καμία περίπτωση βεβαίως δεν μπορεί αυτό να περιοριστεί στο εξάμεινο μιας Ευρωπαϊκής Προεδρίας. Θα πρέπει, όπως και όλα τα άλλα θέματα διακυβέρνησης, να ειδωθούν πολύ πιο διαχρονικά όπως ο κύριος Μόντι, τότε επίτροπος, ε, μιλώντας ε, το 2009 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις συστάσεις του, στην εκθεσή του, είχε κάνει μια τέτοια πολύ εμπεριστατωμένη πρόταση Ξέρω ότι οι προτάσεις αυτές ε, υποστηρίζονται από όλες τις πολιτικές ομάδες. Αυτές είναι οι ενδείξεις που έχουμε. Είμαι λοιπόν αισιόδοξο και σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω γιατί δεν μπορούμε να σβήσουμε αυτό το φως πάνω από τα διαφάνειες, αλλά τέλος πάντων, επειδή θα έχουμε παρουσιάσεις, ε, καλό θα ήταν οι ε, οι υπηρεσίες της Επιτροπής μας να μας ε, βοηθήσουν με μια πολύ απλή έτσι, με ένα πολύ απλό μηχανισμό για να μπορούμε να σβήνουμε το φως πάνω από, τη... από τις διαφάνειες. Τέλος πάντων, να ανάψουμε τώρα τα φώτα τα κανονικά. Ήταν πολύ χρήσιμη παρουσίασή σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δουλειά σας. Είναι πολύ σημαντική η πολιτική αυτή έκθεση για την Επιτροπή μας και ευθυγραμμίζεται και με τις συζητήσεις που είχαμε και προηγουμένως. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την πολύ απλή ξεκαθαρή προσέγγισή σας. Ας ακούσουμε τώρα τους σκιώδεις. Ο πρώτος είναι ο κύριος Κοφεράτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Σβάπ, Αγαπητέ συνάδελφοι, σας ευχαριστώ που παρουσιάσατε με τον τρόπο που το κάνατε αυτό το θέμα. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Σφάπ κυρίως γιατί ανέφερε ένα πολύπλοκο και λεπτό ζήτημα και είπε ότι δεν έχει την πρόθεση να περιοριστεί απλά σε μια άσκηση προσαρμογής, αλλά να αλλάξει τα πράγματα με ριζικό τρόπο. Πρέπει να αλλάξουμε την προσέγγιση, να προσπαθήσουμε να προτείνουμε μια προσέγγιση που θα δώσει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό το ζήτημα της ενισχύσεως, κάτι βέβαια που είναι ήδη σημαντικό και για την Επιτροπή μας και για το Κοινοβούλιο ευρύτερα. Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις σας, αγαπητοί συνάδελφε, και αναφέρουμε στο πώς μπορούμε να βελτιώσουμε και να ενισχύσουμε τις ε, σχέσεις ε, μεταξύ νομιού και κρατών μελών. Αυτή τη στιγμή όλοι θέλουμε να αναγνωριστεί η λειτουργία και ο ρόλος της ε, εσωτερικής αγοράς. Όμως τα μέτρα που περιλαμβάνουν είναι σε εθνικό επίπεδο είναι μετροπαθή και γι' αυτό δεν έχουν και την αποτελεσματικότητα που θα θέλαμε. Και θα πρέπει να γίνει μια ανάλυση, όχι ποσοτική κάθε χρόνο, αλλά ποιοτική. Ποιοτική ανάλυση των διατάξεων που έχουν εγκριθεί στον τομέα της εσωτερικής αγοράς. Η διαδικασία η παραβάση δεν αρκεί. Πρέπει να παρακολουθούμε την εφαρμογή των αποφάσεων. Πώς εφαρμόστηκαν τι προβλήματα ενδεχομένως προέκυψαν, πώς μπορούμε να διορθώσουμε τις τρευλώσεις που παρουσιάζονται ενδεχομένως. Καλό θα ήταν λοιπόν να κάνουμε όσο το δυνατόν πιο νωρίς τις διορθώσεις και να επιβάλλουμε και ε, τις κυρώσεις που απαιτούνται. Πρέπει να κάνουμε να βγούμε προς τα μπροστά και να καταθέσουμε μια νομοθετική πρόταση ώστε ό,τι από τη εσωτερική αγορά να ενταχθεί στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Να είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα τη οικονομική πολιτική όπω αυτή. Θα αποφασιστεί βασιζόμενη βέβαια σε ζητήματα τα οποία καλούμαστε εδώ να εξετάσουμε. Καλή προσέγγιση και πρέπει να την υποστηρίξουμε. Θα πρέπει να συζητήσουμε τα τεχνικά σημεία της ε, έκθεσης και εδώ αναφέρομαι στο άρθρο 27 της συνθήκης, τη νομική βάση στις περιπτώσεις αυτές που είναι αρκετά συγκεκριμένη, αλλά δεν θα πρέπει να σταματήσουμε μπροστά στα τεχνικά εμπόδια. Στόχος μας θα πρέπει να είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως, να είμαστε ιδιαίτερα φιλόδοξοι, αλλά να φανούμε και στο ύψος των σημερινών περιστάσεων και συγκυριών. Ιδάλλως θα ασχοληθώ με ζητήσιμα που είναι σημαντικότατα με την ευρωπαϊκή οικονομία και τελικά δεν αναγνωρίζονται ποτέ επισήμως ως προτεραιότητες. Και μιλάμε για επίσημη αναγνώριση και ως προς την ουσία. Έπειτα θα υπάρξουν και άλλα θέματα που θα πρέπει να ενσωματωθούν λόγου χάρη, η βιομηχανική πολιτική, ως προτεραιότητα που θα πρέπει να αναλυθεί δράση. Θα το συζητήσουμε και με τον Επίτροπο όταν θα τον ε, δούμε. Πάντως νομίζω ο πυρήνας της ε, έκθεσης ε, ΣΦΑΜ είναι αυτός που προανέφερα. Και θα πρέπει να είμαστε πιστικοί στην προσέγγιση μα. Ο κύριο Σφαμπ στην έκθεση του θα πρέπει να κάνει κάποια μνήμα και για το σύνολο των κανόνων των, του Single Market 2, τη ενιαία αγορά 2 δηλαδή, και να δούμε κατά πόσον θα μπορούσαμε να επικεντρωθούμε περισσότερο στο σημείο της προσαρμογής που τόσο πολύ αναμένεται και να δούμε κατά πόσον η ενιαία αγορά θα πρέπει να προσαρμόζεται και σε άλλου είδους συγκυρίες με ανάλογη διατάξεις. Σας ευχαριστώ κύριε Κοφεράτη, ο κύριος Μάντερς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Αντρέας είναι ένα θέμα πολιτικό. Και κάποιες φορές ε, νιώθω ως τεχνοκράτησα όταν συστάμε για κάποια ζητήματα που είναι πάρα πολύ δύσκολο να μεταδώσουμε ε, τα μηνύματα στη κοινωνία. Η ενιαία αγορά είναι ίσως η πιο επιτυχημένη πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο την τελευταία 20 ετία. Επισήμανε ο Αντρέας ότι το 2011 είχαμε 922 διαδικασίες επί παραβάσει διότι τα κράτη-μέλη είχαν υλοποιήσει ή ερμηνεύσει την νομοθεσία κατά το δοκούν. Σταχυολόγησαν δηλαδή τα πράγματα και ενέκριναν μόνο τα μέτρα που τους ε, άρεσαν. Συμφωνώ ότι πρέπει να γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Θα το δούμε. Αφού κάνουμε όμως την ανάλυση που πρέπει να γίνει, πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την εφαρμογή. Πώς εφαρμόζουμε την νομοθεσία. Μπορεί να πρέπει τα πράγματα να γίνονται καλύτερα όχι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά σε επίπεδο κρατών μελών. Συμφωνώ με αυτέ τι συστάσει προ τα κράτη-μέλη, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν διαφορετικέ προσεγγίσεις στα κράτη-μέλη. Με ικανοποιεί ιδιαίτερα κύριε Πρόεδρε που βλέπω ότι τελικά πίεσα και κατάφερα ο Αντρέας να βάλει στο κείμενο ότι οι κανονισμοί είναι καλύτερα από τις οδηγίες. Χρόνια το λέω. Και είναι η μόνη λύση νομίζω για να ξεπεράσουμε κάποια προβλήματα που σχετίζονται με την οικονομική νομοθεσία και την εφαρμογή της. Υπάρχει όμως και ένα ακόμη ζήτημα που ετέθηκε, αυτό είναι η παρακολούθηση και η εφαρμογή. Ίσως θα έπρεπε να υπάρχει ένα σύστημα, ένα είδο δικτύου ε, κάποιων που ελέγχουν την εφαρμογή και κοινοποιούν τα σχετικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για να αποφύγουμε βέβαια τις δυσκολίες και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει όταν τα θα πρέπει όταν προετοιμάζουμε την νομοθεσία να εμπλέκουμε σε αρκετά πρώιμη φάση και τα εθνικά κοινοβούλια για να έχουμε τη δική τους ε, συνεισφορά, έτσι ώστε η νομοθεσία που θα εγκρίνουμε θα είναι μια νομοθεσία που θα μπορούν να την εγκρίνουν και τα εθνικά κοινοβούλια και τα κράτη-μέλη. Γιατί τελικά αν ε, μπουν στο τελευταίο στάδιο της δικασίας τα, κράτη, τα κοινοβούλια τα εθνικά, τελικά έχουν 27 διαφορετικούς τρόπους εφαρμογής νομοθεσίας επευκαιρία της 20 από επαιτίου αποτέλεση τη εσωτερική αγοράς ζήτησα από διάφορες ε, μικρομεσαίε επιχειρήσεις να μου δώσουν σύντομα τις απόψεις τους για το πώς πιστεύουν ότι μπορεί να βελτιωθεί η εσωτερική αγορά. Και την καθημερινότητά τους. Ίσως η Κομισιόν θα μπορούσε ίσως να στείλει σε όλες τις ΜΜΕ αυτή τη, ίσως, ε, την ερώτηση. Να πει δηλαδή στις ΜΜΕ, πείτε μου με 25 λέξεις τι πρέπει να βελτιωθεί στην εσωτερική αγορά. Ή θα μπορούσαμε να διοργανώσουμε και μια ακρόαση για να έχουμε μια ξεκαθαρή Τα πράγματα πρέπει να βελτιωθούν. Εντάξει, πώς όμως. Και πρέπει να σταθμίσουμε βέβαια και τα πολιτικά ζητήματα. Αυτό που μου άρεσε με την παρουσίαση του Αντρέα είναι αυτό που τόνισε, ότι λείπει η επικοινωνία. Τα τελευταία 20 χρόνια δεν έχουμε μεταδώσει προ τα έξω τι σημαίνει για του ευρωπαίου πολίτε η εσωτερική αγορά, τι σημαίνει για την Ευρώπη συνολικά η εσωτερική αγορά. Και νομίζω ότι πρέπει να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφο στον τομέα τη επικοινωνία. Και έχω μια ερώτηση προ τον εισηγητή. Λέει στο σημείο ε, την πολιτική αξιολόγηση. Τι θα πει η political evaluation Ευχαριστώ πάντως τον Αντρέας. Και όταν έχουμε αυτή την πολιτική αξιολόγηση το Δεκέμβριο, στο Λίωνο, ελπίζω να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο πολιτική προσέγγιση, όχι μόνο την τεχνοκρατική, σε ό,τι την οικονομική νομοθεσία. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ για τις πολύ σαφείς σας ιδέες. και για πρώτη φορά δεν μπήκε αυτή η διάκριση κανονισμό σε οδηγία στη... στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου. Κυρία Ρούλε έχει κάτσει στο Προεδρείο γιατί θα τη δώσω τη σκητάλη διότι πρέπει να συναντήσω τον υποψήφιο επίτροπο. σα πάω, θα αλλάζουμε τη σκητάλη γιατί θα μπαινοβγαίνω εδώ. τέλο πάντων ε, η κυρία Ρούλε έχει το λόγο και ότι εισηγήτρια για αυτό το ζήτημα. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Σβάπ. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα της ενέας αγοράς με στρατηγικό τρόπο. Και φυσικά όσον αφορά την υλοποίηση υπάρχουν πολλά που θα έπρεπε να γίνουν με καλύτερο τρόπο. Εμείς ε, βεβαίως στη Γερμανία έχουμε την αξιολόγησή μας για το ποιες είναι οι χώρες που ε, μεταφέρουν με τον καλύτερο τρόπο και υλοποιούν με τον καλύτερο τρόπο τις ευρωπαϊκές ε, ε, οδηγίες. Απ' την άλλη μεριά, αν συγκρίνει κανείς ε, αυτά που γίνονται στη χώρα του με άλλες περιπτώσεις σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη διαπιστώνει ότι δεν είναι πάντα εξαιρετική η κατάσταση. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η συγκριτική αξιολόγηση και να δούμε ε, που υπάρχουν κενά και αδυναμίες όχι μόνο στην μεταφορά στο εθνικό δίκαιο αλλά και γενικότερα στην νομοθεσία. Να γίνει δηλαδή μια αξιολόγηση, να δούμε πού υπάρχουν ακόμα κενά και αδυναμίες και πού μπορούμε να καλύψουμε και να ε, ενισχύσουμε, να συμπληρώσουμε. Καταλαβαίνω πολύ καλά ποιο είναι το ζητούμενο εδώ. Ποια είναι η πρόκληση. Υπάρχουν προβλήματα μεταφοράς, ε, υλοποίησης και στην ε, μεταφορά κανονισμών, όχι μόνο για τις οδηγίες. Και εκεί υπάρχουν διαδικασίες επί παραβάση. Όταν μιλάμε για κανονισμούς, πολλές φορές βλέπουμε ότι τα κείμενα αυτά δεν μπαίνουν τόσο πολύ σε λεπτομέρειες, σε βάθος. Πρόκειται κατά κάποιο τρόπο για ένα κείμενο πλαίσιο, το οποίο δεν μπαίνει τόσο πολύ σε λεπτομέρειες. Αν πάρει κανείς παραδείγματος χάρη τις 214 ε, σελίδες του κανονισμού για την ανάθεση και τις παραχωρήσεις διαπιστώνει ότι είναι αδύνατο να μπει κανείς σε κάτι το πιο συγκεκριμένο. Θα πρέπει λοιπόν ίσως κάποια στιγμή να δούμε ποιο είναι το γενικό πνεύμα αυτού του κείμενου πλαισίου, αυτού του κείμενου κανονισμού, το οποίο επαναλαμβάνω δεν μπαίνει στις λεπτομέρειες, δεν εμβαθύνει όπως ε, πολλές φορές κάποια κείμενα οδηγίες. Εκεί λοιπόν σε αυτή τη σύγκριση δημιουργούνται δυσκολίες και αμφιβολίες και γι' αυτό και εγώ πολλές φορές αμφιβάλλω για τις ε, βεβαιότητές μας. Πρόεδρος. Χαίρομαι που μπήκαμε στην καρδιά του θέματος. Λίγα σχόλια τώρα και από μένα. Η κυρία Μακλάρκιν είναι η σκιώδη μα, αλλά ε, το, παρα, το παρακολουθώ και εγώ πολύ στενά το θέμα, διότι στην διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, όπου έπρεπε να, να περασπιστώ τη θέση τη Επιτροπή μα, Εκεί συμφωνήθηκε να έχουμε νομοθετική έκθεση. Κάτι που βρήκε σύμφωνο στους περισσότερους συναδέλφους. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα ε, ανακύψει το Νοέμβριο και τότε θα επέρασπω στο τη θέση της Επιτροπής μας. Κατά πρώτον, νομίζω ότι είναι ζωτική σημασία στο ζήτημα. Θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε με μεγάλη προσοχή. Η πράξη για την έννοια αγορά ήταν μια προσπάθεια εντατική όλων των κοινοβουλευτικών επιτροπών και η συνεργασία μα ήταν ε, πραγματικά αποδοτική. Αυτό είναι που πρέπει να συνεχιστεί ως κάτι που πρέπει να συνεχιστεί ω προσπάθεια. Διότι μιλάμε για ζητήματα που θα απασχολήσουν ταυτόχρονα πολλέ διαφορετικέ επιτροπέ. Θα πρέπει λοιπόν το Κοινοβούλιο να είναι πιο αποτελεσματικό στην εργασία του και στι αποκρίσει του στο όλο θέμα. Στην ενιαία αγορά και τον κύκλο αυτών των νομοθετικών μέτρων θα πρέπει να αναλάβουν τι υποχρεώσει του, όλε οι επιτροπέ. Για την ενιαία πράξη 2 θα πρέπει λόγω χάρη να δοθεί μια προτεραιότητα στα προγράμματα για τι μεταφορέ. Αυτό το έχουμε ξανασυζητήσει στην Επιτροπή μα. Οι μεταφορέ, οι ουσιαστικέ πραγματικέ μεταφορέ που θα καλύψουν τι ανάγκε βιωσιμότητα και τη ανταγωνιστικότητα σε μια οικονομία που γνωρίζει όλες αυτές τις αλλαγές είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει και να ε, ενταχθεί στο γενικότερο πλαίσιο της λογιστικής μας για την ενιαία αγορά. Όλοι αυτοί οι τομείς είναι τομείς όπου θα πρέπει να έχουμε αντατικότερη συνεργασία και με τα εθνικά κοινοβούλια. Είχαμε κάποιες επιτυχείς ε, συζητήσεις και συνομιλίες με τα εθνικά κοινοβούλια για θέματα όπως τα δικαιώματα των καταναλωτών, κάτι που απασχολεί πολύ σοβαρά τους εθνικούς βουλευτές αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει τέτοια, τέτοιο ενδιαφέρον και να συναρπάζονται τα εθνικά κοινοβούλια από την ευρύτερη σημασία τη ενιαία αγορά. Είναι πολύ σημαντικό όμω. Πρέπει να υπερασπιστούμε την σημασία τη ενιαία αγορά για την δημιουργία θέσεων απασχόληση, για τα συστήματα κοινωνική πρόνοια. Είναι ύψη τη σημασία. Αλλά επισκιάζεται από άλλε προτεραιότητε, ιδίω σε καιρού οικονομική ύφεση. Είναι λοιπόν ένα πολιτικό μήνυμα αυτό που πρέπει να περάσει. Δεύτερη παρατήρηση και εδώ θέλω να επενέσω την ε, συγκίτρια για το έργο της και αυτό προσπαθεί να κάνει και η κυρία Μακλάρκη είναι να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην πραγματική, την ουσιαστική μεταφορά της νομοθεσίας. Το τι ζητήματα ανακύπτουν από την διαδικασία μεταφοράς είναι κάτι που επίσης πρέπει να μας απασχολήσει. Αυτό νομίζω το λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη ο κύριος Φαμπ. Αλλά θα πρέπει να ενδυναμωθεί και η διαδικασία ε, της ενδελεχούς αναθεώρησης των, της ισχύουσας νομοθεσίας. Πρέπει να βελτιωθεί και η ποιότητα της νομοθεσίας. Αυτό είναι κάτι το που ήδη το συζητάμε εδώ και καιρό. Όμως και η Επιτροπή στην μελέτη αντικτύπου της κατέληξε στο συμπέρασμα και μας είπε και παραπονέθηκε ότι δεν αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις τους οι αρχές των κρατών μελών για το σύστημα μεταφοράς της νομοθεσίας ειδικά. Η νομοθεσία πρέπει να σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο που να είναι απλό και αποτελεσματικό το να τη μεταφέρει κανείς. Να είναι και εύληπτη. Αυτό αληθεύει και από τη σκοπιά του κυρίου Μάντερ και των θεμάτων που μα έθεσε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την καλύτερη νομοθεσία. Και οι μηχανισμοί επιβολής είναι σημαντικοί. Όπως γνωρίζουμε από τις διαρκείς εκκλήσεις μας για τη βελτίωση της παρακολούθησης τη αγορά και των μηχανισμών αυτών, κάτι που θα μας απασχολήσει και του χρόνου, είναι ότι με τα κονδύλια που διατίθενται είναι δύσκολο να πείσουμε τα κράτη-μέλη να κάνουν μεγαλύτερε επενδύσει στην παρακολούθηση τη αγορά. Ιδίω για τη συλλογή περισσότερων πληροφοριών λόγω χάρη και στοιχείων. Σε κάποιε περιπτώσει χρειάζεται να συμμετάσχουν περισσότερο και οι επιχειρήσει, παρέχοντα περισσότερε πληροφορίε. Εκεί που εντοπίζουν λόγω χάρη προβλήματα και δυσκολίε. Έχουν πληροφορίε. Απλώς δεν τις μοιράζονται αρκετά μαζί μας. Θα πρέπει να είμαστε τόσο επινοητικοί ώστε να εξεύρουμε τρόπους για να γίνει η ενιαία αγορά και οι πληροφορίες που την αφορούν πραγματικά ε, προτεραιότητα. Μέρος όλη αυτής τη εργασία θα είναι να πιέσουμε τα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν αυτό που διαρκώς ε, ζητούμε. Να συνενώσουν τι υπηρεσίε του σε συλλογές πληροφοριών για την ενιαία αγορά. Αυτό είναι πραγματική προτεραιότητα. Όπως το it, το go, το ενία σημεία επαφή, Όλα αυτά που χρησιμοποιούν στοιχεία και πληροφορίες για την ενία αγορά θα πρέπει να ε, καταλήγουν σε ένα σημείο επαφής οι πολίτε, οι καταναλωτέ που αντιμετωπίζουν προβλήματα, κάτι που συζητήσαμε ήδη το πρωί, το ακούσαμε, ή όσοι παρέχουν αγαθά ή υπηρεσίε, δεν ξέρουν πού να αποταθούν. Αυτό και οι πολίτες το χρειάζονται και από την πλευρά των κυβερνήσεων είναι αναγκαίο. Όλοι λένε χρειαζόμαστε ένα ενιαίο σημείο επαφή, ιδίω στην όλη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Πρέπει κάποιο να ξέρει που να απευθυνθεί. Πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη να ε, δίνουν τι προσπάθειέ του, να μα δίνουν περισσότερε δομημένε, διαρθρωμένε και χρήσιμε πληροφορίε για την ενιαία αγορά και για την υλοποίηση τη νομοθεσία. Είναι ρόλο αυτό και των σημείων επαφή. Πρέπει να βελτιώσουμε λοιπόν την πολιτική διάσταση του θέματος και η ετήσια έκθεση για την ενοποίηση της, αγορές, της αγοράς είναι σημαντικό. Ναι, και οι μικρομεσαίες επιχειρήσει εδώ μπορούν να συμμετάσχουν και από αυτό που είπα και για την ενοποίηση τη νομοθεσία είναι σημαντικό. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσει πρέπει να συμμετέχουν. Και θα επιμείνω στο θέμα αυτό στην όλη συζήτηση όπως επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει την υλοποίηση να τη δούμε όχι μόνο μέσω της δεύτερης πράξης για την ενιαία αγορά, αλλά και των μέτρων της πρώτης πράξης για την ενιαία αγορά που ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Τα επαγγελματικά προσόντα λόγου χάρη. Κάτι που ελπίζουμε ότι θα ολοκληρωθεί το αργότερο φέτος ή στο πρώτο εξάμεινο της επόμενης χρονιάς. Ή το τι συμβαίνει με την ψηφιακή οικονομία και την τρίτη δέσμη μέτρων για τον τομέα αυτό. Νομίζω λοιπόν η βάση που έχουμε είναι πολύ καλή, αλλά και η κυρία Μακλάρκιν και εγώ θα συμβάλλουμε όσο πιο επιδημιουργικά μπορούμε στην επεξεργασία αυτή τη πρόταση. Υπάρχει κάποιο συνάδελφο που θέλει το λόγο, κυρία Τούν. Κάποιος άλλο. Ωραία, κυρία Τούνεν Χόνστα, είναι το λόγο και σε λίγο θα πρέπει να φύγω για τη συνάντησή μου. This is an extremely important Είναι πάρα πολύ σημαντικό το σύντημα αυτό. Ξεκολουθεί όμως να υπάρχει εξή κατάσταση. Η νέα αγορά αντιμετωπίζεται από τα κράτη-μέλη. Σαν να μην είχαν την ευθύνη αυτά. Σαν να είμαστε εμείς εδώ υπεύθυνοι για την ενιαία αγορά και όχι τα κράτη-μέλη. Αυτό το ακούμε συνεχώς, ε, εσείς, εμείς κτλ. Κάτι άλλο, όπως είπαν και οι συνάδελφοι. τα μηνύματα τα οποία ε, στέλνει η Κομισιόν, ότι δηλαδή θα πρέπει οι κυβερνήσεις να συμμετέχουν ε, περισσότερο, είναι πάρα πολύ αδύναμα και όχι μόνο κυβερνήσεις και άλλα, ε, άλλοι κύκλοι. Μίλησε ο κύριος Μάντρες για διαβουλεύσεις. Αυτό είναι ένα σπονοκέφαλος για όλους μας και όχι μόνο. Εγώ συχνά έχω την εντύπωση συγγνώμη που τα λέω έτσι, ομάτα πράγματα, σαν η Κομισιόν να κάνει ότι ε, ζητά τη συμμετοχή άλλων κύκλων, κάτι όμως που τελικά δεν ισχύει, γιατί δεν τους προσκαλεί τους κύκλους αυτούς ε, στις διαβουλεύσεις, γιατί κανείς δεν γνωρίζει τίποτα για τις διαβουλεύσεις αυτές τελικά, δεν συμμετέχει κανένας. Ή αν ε, υπάρχουν κάποια έγγραφα, αυτά είναι είτε μόνο στα αγγλικά είτε σε τρεις γλώσσες. Ποτέ σχεδόν σε όλες τις επίσημες γλώσσες και είναι και ιδιαίτερα πολύπλοκα τα ζητήματα αυτά. Άρα οι παραλήπτες συχνά δεν τα καταλαβαίνουν. Ο Ανδρέας ανέφερε σε ένα ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό. Με την Κομισιόν και εκεί οι συζητήσεις μας είναι πάρα πολύ δύσκολες για την ευθύνη. Ποιος έχει την ευθύνη πρέπει να μιλήσουμε με τις ΓΔ Μάρκτ και ΣΑΝΚΟ πιο ειλικρινά και να δούμε πώς μπορούμε να ε, δώσουμε σάρκα και οστά σε αυτή την προθυμία. Πρέπει σίγουρα την ευθύνη να την έχει η Κομισιόν, αλλά έχουμε και εμείς ευθύνη να πιέσουμε. Ένα σημείο πρέπει να έρχουμε. Έχω δει κι εγώ πόσο δύσκολο είναι. Παραδείγματο χάρη, όταν διαπραγματευθήκαμε την ε, επίλυση διαφορών online, αυτό είναι κάτι που θα ήθελα να μπει σε αυτή τη ε, διεύθυνση, το ενιαίο σημείο επαφή, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να πείσουμε του φίλους μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσουν το ένα αυτό σημείο επαφή. Που υπάρχει τελικά το Europe και δεν το χρησιμοποιούμε. Σε ό,τι αφορά τα εθνικά κοινοβούλια. Νομίζω ότι οι εθνικέ ε, διοικήσει και άλλοι κύκλοι στα κρατημέλη δεν συμμετέχουν αρκετά και κάτι άλλο το οποίο θα ενίσχυε είναι ο ρόλος των φόρουμ ε, για την ενιαία αγορά. Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Να χρησιμοποιήσει περισσότερα τα κοινωνικά μέσα ε, δικτύωσης, το web streaming, όπως τελευταία φορά όταν ξεκίνησε το φόρουμ για την ενιαία αγορά εδώ. Ώστε η ενιαία αγορά να είναι ένα ζήτημα όχι μόνο για αυτούς που είναι εδώ στις Βρυξέλλες, αλλά σε όλα τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Αν κατάλαβα καλά, η Επιτροπή δεν είναι προετοιμασμένη, άρα δεν θέλει να πάρει το λόγο. Θέλετε? Όχι. Όχι, δεν θέλετε να αντιδράσετε. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει θέμα. Ο εισηγητής συμπερασματικά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν ευχαριστώ όλους για τα πολύ επικοδομητικά και τα πάρα πολύ χρήσιμα ε, σχόλιά τους. Πάρα πολύ χρήσιμα και πιστεύω πραγματικά ότι εδώ μπορεί να υπάρξει συζήτηση και απόφαση μόνο σε πολιτικό επίπεδο. Ελπίζω να το κάνουμε. Ελπίζω την επόμενη φορά η Επιτροπή θα στηρίξει αυτήν την ε, πρόταση και καταρχήν θα συμμετάσχει και στην συζήτηση. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια από τα σημεία. Ευχαριστώ τον κύριο Κοφεράτη για τη στήριξή του, για τα σχόλιά του. Τον ευχαριστώ πολύ γιατί θεωρώ πραγματικά ότι πέρα από τα τεχνικά προσκόμματα και δυσκολίες θα πρέπει να μπούμε στην ουσία. Και ελπίζω ότι θα το πετύχουμε αυτό. Είμαι ανοιχτό σε κάθε επικοδομητική πρόταση. Ξέραμε ε, από την αρχή ότι το θέμα αυτό είναι φορτισμένο. Και βεβαίως η ενιαία πράξη 2 είναι κάτι που μας έχει οδηγήσει σε τοποθετήσεις. Το ίδιο θα κάνουμε και για την ενιαία πράξη 3 προφανώς. Εγώ μίλησα για το εξάμεινο της Προεδρίας, για αυτό το εξάμεινο το οποίο θέλουμε να οργανώσουμε με συγκεκριμένες προθεσμίες και ημερομηνίες. Θα ήθελα να σας πω ότι για την ενιαία πράξη 2 θα υπάρξει μια ξεχωριστή παρουσίαση, ένα ξεχωριστό κεφάλαιο και ότι το ευρωπαϊκό αυτό εξάμεινο σαφώς και θα ενσωματωθεί στην πρότασή μας έτσι ώστε όλοι να μπορέσουν να κάνουν προτάσεις και να συμμετάσχουν. Σε καμία περίπτωση δεν έχει νόημα να μην υπάρχει συμμετοχή όλων των ε, ενδιαφερομένων σε αυτήν την διαδικασία. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι και η ΚΟΖΑΚ, δηλαδή η συνάντηση των Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων, Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και οι πρόεδροι των κοινοβουλίων με κάλεσαν στη Λευκοσία στην τελευταία τους συνεδρίαση για να παρουσιάσω τις σκέψεις και τις προτάσεις μας. Βεβαίως μπορεί κανείς να πει ότι εδώ υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα επικοινωνίας ενημέρωσης και αυτό ιδιαίτερα όταν υπάρχουν πολύ σημαντικές πολιτικές ε, αποφάσεις που διακυβεύονται. Γι' αυτό και είπα προηγουμένως συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων σε όλα τα επίπεδα γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα θετικό πνεύμα. Να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή όχι μόνο για θέματα μακροοικονομικής ανάλυσης αλλά, αλλά παράλληλα με τους συναδέλφους όλων των αρμόδιων επιτροπών που εμπλέκονται για την υλοποίηση αυτών των εκάστοτε οδηγιών, είναι μια μοναδική ευκαιρία να αυξήσουμε τις δυνατότητες επιτυχίας. Όσον αφορά λοιπόν το θέμα της υλοποίησης νομοθετικών κειμένων που αφορούν την ενιαία αγορά, αυτό όπως ε, καταλαβαίνετε προσκρούει σήμερα στι οικονομικέ δυσκολίε που αντιμετωπίζουν κάποιε χώρε. Καταλαβαίνουμε ότι μια χώρα που σήμερα βρίσκεται εν μέσω οικονομικών δυσκολιών ε, που αναγκάζεται να περάσει κείμενα ε, επιγόντως ε, τα οποία αφορούν αυτή την οικονομική κατάσταση, σίγουρα θα επιβραδύνει σημαντικά την μεταφορά κάποιων νομοθετικών κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την ενιαία αγορά σε σχέση με μια άλλη χώρα όπου υπάρχει μια ε, σταθερή διακυβέρνηση και κυβερνητική διαδικασία, νομοθετική, κοινοβουλευτική διαδικασία. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να θέσουμε κάποιες ε, προτεραιότητες οι οποίες να ισχύουν για όλους, λαμβάνοντας βεβαίως υπόψη της ιδιαιτερότητας. Άκουσα πολύ προσεκτικά και αυτό που είπε ο κύριος Μάντες όσον αφορά την πληροφόρηση, την ενημέρωση. Εδώ μπορούμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα. Πιστεύω επίσης ότι είναι πολύ ορθό αυτό που είπατε, κυρία Πρόεδρε, για, τις, για τους κανονισμούς. Όντως θα πρέπει εδώ να εξετάσουμε και το θέμα αυτό. Κύριε Μάντελς, μιλήσατε για την αξιολόγηση, την αξιολόγηση από μακροοικονομικής απόψεως. Ναι, αλλά όχι μόνο αυτός ο τομέας θα πρέπει να αξιολογηθεί. Όταν μιλούμε για ενιαία αγορά, πολλές φορές βλέπουμε ότι η μεταφορά και η υλοποίηση γίνεται όχι ολοκληρωμένα. Και η Επιτροπή εδώ βεβαίως πρέπει να παίξει ένα ρόλο επιτήρησης, ελέγχου. Η μακροοικονομική πλευρά σαφώς και θα πρέπει να συνεχίζει να παίζει ένα καθοριστικό ρόλο, αλλά η υλοποίηση όλων των υπόλοιπων καλώνων που αφορούν την ενιαία αγορά και αυτό και αυτή η δραστηριότητα θα πρέπει να γίνει πρωταρχική σημασία. Η κυρία Ρουλίπε και ο κύριος Κοφεράτη ότι βεβαίως ο καθένας μπορεί στην χώρα του να κάνει κάτι. Θα πρέπει να ενημερώσουμε την κοινή γνώμη των χωρών και θα πρέπει από κοινού να υποστηρίξουμε τις απόψεις μας. Και όπως ε, βεβαίως έγινε με την τελευταία, το τελευταίο παράδειγμα για την οδηγή ανάθεση, βλέπετε ότι σε καμία περίπτωση ένα τέτοιο θέμα δεν θα πρέπει να γίνει θέμα εθνικής ε, αντιπαράθεσης είτε αντιπαράθεσης μεταξύ των διαφορετικών εθνικών θέσεων. Βλέπετε επίσης τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλές φορές μεγάλες χώρες όπως πρόσφατα παραδείγματα να ζητήσουν ε, υποστήριξη, βοήθεια. Αυτό πιστεύω θα πρέπει να ρυθμιστεί στην ιδέα και στην πρόταση για το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Η υλοποίηση θα πρέπει να είναι η ίδια, να βασίζεται σε κοινού στόχους. Εμείς εδώ σαν μέλη του Κοινοβουλίου πρέπει να παίξουμε το ρόλο μας. Θα αναφερθώ εδώ σε αυτό που είχε πει ο Επίτροπος Μπόλκενστάιν πριν από χρόνια για την ε, εσωτερική αγορά λέγοντας ότι βρισκόμαστε μέσα σε μία Φεράρι με απεριόριστες δυνατότητες επιτάχυνσης. Είμαστε όμως ακόμα στη δεύτερη ταχύτητα. Δεν έχουμε περάσει στην πραγματική ταχύτητα που μπορεί να πιάσει αυτό το αυτοκίνητο. Ας περάσουμε λοιπόν. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. 12 Νοεμβρίου είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Μπορείτε όμως να υποβάλλετε τροπολογίες και μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου στις 12 υπάρχει... Όχι, δεν υπάρχει ακόμα απόφαση. Θα το αποφασίσουν οι συντονιστές, λέει η Πρόεδρος, αύριο αυτό. Αν αλλάζει η προθεσμία και γίνεται 6 Δεκεμβρίου η ψηφοφορία θα γίνει τον Ιανουάριο 23-24 ε, Ιανουαρίου εδώ στην Επιτροπή και το Φεβρουάριο στην Ολομέλεια. Ωραία, πολύ ωραία. Ολοκληρώσαμε αυτό το σημείο της ημερής σας διάταξης και τώρα περάμε στην επόμενη έκθεση που είναι το θέμα των τελωνίων 2014-2020. Ο κύριος Μπαλτιζάρη έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε μετά την απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων στις 16 Μαΐου 2012, όπου υποστηρίχθηκε η αίτηση διαχωρισμού των δύο προγραμμάτων για τα φορολογία και τα τολενία, μετά την, ε, το επίσημο αίτημα των Επιτροπών ΙΜΚΟ και ΕΚΟΝ τροποποιήθηκε και η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να ληφθεί υπόψη η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Έτσι, στι 29 Αυγούστου εγκρίθηκε τροποποιημένη πρόταση των προγραμμάτων για τα τελωνία 2020 και για τη φορολογία 2020. Και οι δύο επιτροπέ οικονομικών υποθέσεων και προστασία καταναλωτών και εσωτερική αγορά είχαν επισημάνει διάφορε ασάφειε των προγραμμάτων και επισημένοντα τα πλεονεκτήματα του διαχωρισμού των δύο αυτών προγραμμάτων. Βάσει της νέας πρότασης για το νέο δημοσιονομικό πολιετές πλαίσιο, ο κανονισμός για τα τελωνία για τα τελωνία μέχρι το 2020 προβλέπει ένα κονδύλιο 250 εκατομμυρίων ευρώ ως το, για το επόμενο επταετές ε, χρονικό διάστημα. Έτσι λοιπόν το αρχικό πρόγραμμα που τώρα έχει διαιρεθεί σε δύο είναι κάτι που μας ικανοποιεί ιδιαίτερα, όπως επίσης και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως προτείνεται. Θεωρώ σημαντικό βεβαίω να υποβληθούν κάποιε τροπολογίε και να γίνουν κάποιε τροποποιήσει στο κείμενο, τι οποίε αυτή τη στιγμή εξετάζουμε. Για λόγου νομική αφήνεια και καθαρότητα, οι προτεραιότητέ μα θα πρέπει να μετατραπούν σε συγκεκριμένου στόχου στο άρθρο 6. Και θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο ίδιο το σώμα του κανονισμού. Επίσης, σημαντική ήταν η οικονομική προοικοδότηση του προγράμματος. Αυτό βέβαια αφού ολοκληρωθούν συζητήσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο θα το δούμε. Και επίσης θα πρέπει να υπάρξει συμβολή για την διατήρηση και τον εξοπλισμό για το σύστημα πληροφορικής και συγκέντρωσης πληροφοριών. Δεδομένου και του προηγούμενου του προηγούμενου προγράμματος για τα τελωνία, Customs 2013, που προβλεπόταν ένα επίπεδο χρηματοδότησης 75-80%. Θα πρέπει το πρόγραμμα να καλύπτει όχι μόνο τις κοινέ δράσεις για την ανάπτυξη και την καλλιέργεια των ε, δυνατοτήτων υπολογιστών και του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και την ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων. Υπάρχουν ε, στοιχεία τα οποία από τεχνικής άποψης είναι πολύ σημαντικά, όπως η μέτρηση των επιδόσεων και σκόπιμο θα είναι να εκχωρηθούν κάποιες αρμοδιότητες στην Επιτροπή βάσει του άρθρου 290 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι θα μπορεί να χρησιμοποιούνται η, κατεξουσιοδότηση, η κατεξουσιοδότηση πράξης πέραν ε, των όσων θα προτείνει το Κοινοβούλιο και όπως ορίζει βεβαίως η σχετική διάταξη για την εικόνα δρομοδιοτητών στην Επιτροπή. Καλό θα είναι να τονιστεί ότι η Επιτροπή θα καλύψει το κόστος ε, των εξελίξεων που θα επιβληθούν από τις ενωσιακές ε, προσαρμογές και θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην εναρμόνιση και την ε, τυποποίηση των ε, τελωνιακών διαδικασιών. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία. Δεν θα μακρηγορήσω τώρα για το περιεχόμενο της νομοθετικής έκθεσης. Ε, η λογική έκθεση τα αναπτύσσει αυτά διεξοδικά. Ελπίζω απλώς οι συνάδελφοι που είναι παρόντες και αυτοί που απουσιάζουν να κάνουν σχόλια Περιμένω λοιπόν και τη δική του συνεισφορά για να μπορέσει να εμπλουτιστεί η σύνταξη τη έκθεση. Ό,τι αφορά το ίδιο το πρόγραμμα, όριο για την υποβολή τροπολογιών ορίζεται στι 12 Νοεμβρίου. Ω τότε είμαι στη διάθεσή σα. Ευπρόσδεκτα όλα τα σχόλια και όλε οι παρατηρήσει. Σα ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κοφεράτη είχε στήσει το λόγο, αλλά θα ήθελα να δώσω το λόγο καταρχάς στον κύριο Σμιτ γιατί θέλει να φύγει. Συμφωνείτε κύριε Κοφεράτη να δώσω πριν από εσάς το λόγο στον κύριο Σμιτ. Ωραία. Κύριο Σμιτ, να ευχαριστήσω καταρχά τον κύριο Κοφεράτη. Ξέρετε, πρέπει να είμαι σε 10 λεπτά σε μια άλλη επιτροπή και ζητώ συγγνώμη. Αυτά τα προβλήματα έχει κανείς όταν είναι σε μικρή ομάδα. Εσείς δεν το έχετε ποτέ φαντάζομαι αντιμετωπίσει, αλλά εμείς το αντιμετωπίζουμε. Λοιπόν, είναι πολύ καλή πρόταση και συγχαίρω και ευχαριστώ τον εισηγητή για τις εισαγωγικέ του παρατηρήσεις. Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα 27 κράτη-μέλη, αλλά και για τα άλλα βέβαια. Ε, θέλουμε να εφαρμοστεί. Σύντομα θα είμαστε 28. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως έχουμε συζητήσει και κατά το παρελθόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ένα νέο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών και εξεχρονισμένο ε, σύστημα για τα τελωνία. Είτε το ότι είναι κοινοτική αρμοδιότητα είτε γενικώ. Θέλουμε να είναι αρμονισμένο το σύστημα. Το πρόβλημα βέβαια θα μπορούσε να είναι το κόστο. Το έχουμε ξανασυζητήσει και το ανέφερε και η τα κράτη-μέλη, κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα συμφωνήσουν ότι είναι αρμόδια για τη χρηματοδότηση του νέου συστήματος ε, πληροφοριών, η IS. Προς το παρόν, μάλιστα, δεν ξέρουν καν γιατί είναι υπεύθυνοι ή αρμόδιοι. Σίγουρα για τη χρηματοδότηση, πάντως, ευρωπαϊκή. Θέλω να δούμε και ποια θα είναι η αράξη προτεραιοτήτων και τι θα γίνει με την κοινή διαχείριση, Η κοινή τελωνική διαχείριση. Είναι ένα από τα πολύ σημαντικά ζητήματα. Η Κομισιόν λέει ότι κάποια ή όλα. Some or all. Ότι αυτό αφορά κάποια ή όλα τα κράτη-μέλη. Τι εννοείται ακριβώ, δεν θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό για όλα τα κρατη Τώρα η υλοποίηση λέει ότι οδήγησε στη κατάρριση των τελωνικών διατυπώσεων κτλ. Και αυτό οδήγησε σε πολλά πλεονεκτήματα. Ναι, αλλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι και το οργανωμένο έγκλημα χρησιμοποίησε. Εγώ είμαι μέρος της Επιτροπής Κρίμ, όχι crime που τη λένε πολλοί, Επιτροπής Κρίμ. Και ξέρουμε ότι κάθε χρόνο εκατομμύρια δισεκατομμύρια ακόμη ευρώ χάνονται σε αυτό το είδου τα εγκλήματα. Και μια από τις βασικές προτεραιότητες ε, των ε, επιχειρήσεων κατά της απάτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η παράνομη διασυνοριακή διακίνηση αγαθών, εμπορευμάτων. Υπάρχει και μια ομάδα εργασίας του Συμβουλίου και οι όλα προσπαθούν να βελτιώσουν τη διασυνορική συνεργασία. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω ότι θεωρώ πως θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προτεραιότητα σε αυτά τα μέτρα. Και τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να βελτιωθεί η συνεργασία. Με τα χαρά θα συνεργαστώ με τον εισηγητή, του Σκιώδης και ευχαριστώ εκ νέου τον κύριο Κοφεράτη που μου παραχώρησε τον λόγο. Κυρία Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κοφεράτη που παραχώρησε ευγενώς θέση του και να δώσω τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω κι εγώ, όπως είπε ο συνάδελφος Μπαλντασάρε, ότι αυτό που αποσπάσαμε από την Επιτροπή είναι ένα άριστο αποτέλεσμα. Είναι κάτι που το υποστηρίξαμε από την αρχή της συζήτησης, αλλά το αποφεύγανε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή διέρεση του προγράμματος σε δύο τμήματα υπήρχαν στοιχεία, συνιστώσεις του, προγράμμα, του προγράμματος, ε, όπως αρχικά είχε προταθεί, που ήταν βεβαίως αλληλένδετα αλλά, και αλληλένδετες, αλλά επίσης πολύ διακριτά. Οπότε αυτό ήταν ένα θετικό αποτέλεσμα. Και νομίζω καλά έκανε ο συνάδελφος Μπαλτασάρε που σε κάθε περίπτωση προσέθεσε διευκρινιστικές παρατηρήσεις Κάποια σωστά περιλήφθησαν, κάποια άλλα όπως η καταπολέμηση της διαφθοράς νομίζω μπορούν να διευκρινιστούν έτσι περαιτέρω. Θα μπορούσαμε λοιπόν να τα επεξεργαστούμε σε ένα πνεύμα συνεργασίας επικοδομητικό και στη διάρκεια μελέτης του κειμένου. Λόγω χάρη πρέπει να δοθεί έμφαση νομίζω στη συμβολή της πληροφορικής που εξυπηρετεί ως εργαλείο τις τελωνιακές δραστηριότητες. Από την άποψή μου, από τη δική μου τη σκοπιά, πρέπει να τονιστεί ο ρόλος των stakeholder, των ενδιαφερομένων, κάτι που σχολιάζει ο κύριος Μπαλτασάρη στην έκθεσή του, επειδή με μεγαλύτερη, ενεργότερο συμμετοχή, μπορούν να εντοπίσουν, να ε, καταδείξουν τα αρνητικά σημεία των διαδικασιών. Ο ρόλος λοιπόν των stakeholder είναι σημαντικός. Οι γνώσεις τους, οι αρμοδιότητές τους μπορούν να προσδώσουν ποιότητα και γνώση στις τελωνιακές πολιτικές. Νομίζω ότι από τώρα πρέπει να σκεφτούμε ποια θα είναι η σχέση μεταξύ του προγράμματος και των άμεσων και έμεσων δράσεων που μας απασχολούν σε επίπεδο ενιαίας αγοράς, εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να διαρωτηθούμε, χωρίς να καταλήξουμε σε βιαστικά ή πρώιμα συμπεράσματα, εάν το πρόγραμμα φίσκους θα μπορεί να χρηματοδοτήσει και επιπλέον προγράμματα συνεργασίας που συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερος βαθμός διαφάνειας, καλύτερη γνώση των δυναμικών τάσεων της οικονομίας το τι γίνεται με τις διαδρομές που ακολουθούν τα αγαθά, τα εμπορεύματα και οι πολίτες, τα πρόσωπα. Τι διευκολύνει την ε, μετακίνηση των ε, εμπορευμάτων. Θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε το επίπεδο ανταγωνιστικότητα των διαφόρων περιοχών μας και να υπάρξει και ένα επιπλέον στοιχείο συνοχής, εκεί όπου φαίνεται να έχουν γίνει δυναμικά άλματα πρόοδου εδώ να μην παραμελήσουμε και να μην ε, ξεχάσουμε τις ε, θετικέ κινήσεις που έχουν γίνει, αλλά πραγματικά η διαίρεση των δύο προγραμμάτων, ο διαχωρισμό των δύο θεμάτων, μας επιτρέπει να στραφούμε μεγαλύτερο ενδιαφέρον και περισσότερη αποτελεσματικότητα σε συγκεκριμένα στοιχεία του συστήματος πληροφοριών, ώστε να δούμε από μια ευρύτερη σκοπιά την εσωτερική αγορά. Αυτό μπορεί να γίνει με ε, ηρεμία, χωρίς να έχουμε βιαστικά συμπεράσματα και αποφάσεις, διότι νομίζω ότι ο συνάδελφο έχει προσεγγίσει με το σωστό πνεύμα το όλο θέμα. Άλλωστε έχει δείξει μεγάλη διαλεκτικότητα και προθυμία να συνεργαστεί και με τους υπόλοιπους. Äh, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για του ε, πράσινου. Ε, σύντομα θα εκφράσω κάποιες θέσεις. Και εγώ βεβαίω είμαι υπέρ των θέσεων του κυρίου Μπαλτεσάρη. Πάρα πολύ θετικά όλα αυτά που ακούσαμε και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί η Επιτροπή ακολούθησε τις ε, προτάσεις μας. Θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω ότι η Τελωνιακή Ένωση, ο εξυγχρονισμός των τελωνίων είναι κάτι που συνεχίζεται και που ε, σε κάθε περίπτωση, αν δεν υπάρξει αποσαφήνιση της χρηματοδότησης, ε, δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Τι χρειαζόμαστε την Τελωνιακή Ένωση για την ενιαία αγορά και είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως είπε και ο κύριος Σμιτ, να αναρωτηθούμε πώς τα κράτη-μέλη εδώ θα συνεισφέρουν, πώς θα πιέσουμε περισσότερο έτσι ώστε να παίξουν το ρόλο τους εδώ τα κράτη-μέλη και να κάνουν αυτό που καλούνται να κάνουν πώς μπορούμε να ασκήσουμε μια ολοκληρωμένη θα έλεγα πίεση, ενιαία πίεση, έτσι ώστε κάποια πράγματα να γίνουν δεσμευτικά. Χαίρομαι πάντως γιατί το πνεύμα συνεργασίας είναι πολύ καλό. Ε, μέχρι τώρα είχα εντοπίσει τις ε, προτάσεις μου και τις παρατηρήσεις μου στην ε, Τελωνιακή Ένωση. Θα επεκταθώ και στα επόμενα θέματα. Ναι, ο κύριος Μπίλαν. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τις τροπολογίες. Η έκθεση αυτή ουσιαστικά είναι για την, ε, την γνωμοδότηση, μάλλον για την έκθεση Λεγκρίπ. Πριν από έξι εβδομάδε καταθέσαν τι τροπολογίες. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η έκθεση γιατί παρουσιάζει προτεραιότητε, στόχου αλλά και ένα δημοσιομικό πλαίσιο για τα επόμενα χρόνια. Δεν έχω πολλά σχόλια. Διάβασα την πρόταση και βλέπω ότι έχουν συμπεριληφθεί τα σημαντικότερα. Το τελεινικό πρόγραμμα 2013 ήταν πολύ αποτελεσματικό. Ελπίζω και το επόμενο να είναι εξίσου αποτελεσματικό. Να τονίσω όμως ένα σημείο. Συμφωνώ με τον εισηγητή σε ό,τι αφορά την τροπολογία 22 για το δημοσιονομικό πλαίσιο. Συμφωνώ λοιπόν πρέπει να είμαστε ευέλικτοι. Να μην προχωρήσουμε σε πάγωμα πόρων που έχουν ε, που προβλέπονται για αυτό το πρόγραμμα. Στην έκθεση Λεγκρίπ προβλέπονται πολλά μέτρα για τον εξυγχρονισμό των τελωνίων. Πρέπει να αφήσουμε λοιπόν κάποια περιθώρια λιγμών σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση. Πρέπει να είμαστε σε θέση να προσαρμόσουμε τα διάφορα κονδύλια του προπολογισμού. Αυτή ουσιαστικά είναι η σημαντικότερη μου παρατήρηση και ευχαριστώ εκ νέου τον εισηγητή. Θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μπαλτασάρτο και τον κύριο Κομφεράτη για τα σχόλιά τους. Και πρέπει να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει την πρόταση που ακολουθεί τη γραμμή και συνεχίζει το ισχύουν πρόγραμμα που στην ενδιάμεση αναθεώρηση θεωρήθηκε αποτελεσματικό και αποδοτικό. αυτή τη σκοπιά, ω εξακολούθηση αυτών που ήδη κάνουμε, το πρόγραμμα αυτό ε, είναι σημαντικό, αλλά για κάποιε από τι προτάσει που περιλαμβάνονται στα διάφορα σχόλια που ακούστηκαν, πρέπει να κρατήσω κάποιε επιφυλάξει. Εγώ βλέπω τέσσερι κατηγορίε για να απλουστεύσω τα όσα έχω να πω. Πρώτα απ' όλα, η χρηματοδότηση του εξοπλισμού. Στην ενδιάμεση αναθεώρηση. Αξιολόγηση, μάλλον υπήρξαν προτάσεις για νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τον εξοπλισμό. Νέο στοιχείο αυτό. Στη μελέτη αντικτύπου υπήρξε ένα σενάριο για χρηματοδότηση εξοπλισμού μαζί με το πρόγραμμα. Δεν προκρίθηκε όμως αυτό το σενάριο, διότι θα οδηγούσε σε υπέρογγια αύξηση του προπολογισμού και του κονδυλίου. Από την πρόταση του γιατί δεν είναι σαφέ τι είδου εξοπλισμού θα ήθελε να χρηματοδοτούμε. Ο εξοπλισμό από τα κιάλια Ω τα σκάνερ με ακτίνε χ είναι διαφορετικό. Δηλαδή μπορούμε να φτάσουμε από μερικά κατοστάρικα σε εκατομμύρια ευρώ. Δεν έχει εγκριθεί λοιπόν η χρηματοδότηση τέτοιων εξοπλισμών δαπανηρών. Θα είναι πολύ δύσκολο να βρούμε το ανάλογο απόθεμα ή τέλο πάντων τι δυνατότητε χρηματοδότηση εξοπλισμού στα πλαίσια του υπάρχοντος προπολογισμού. Καταλαβαίνουμε από την πλευρά τη Επιτροπή γιατί είναι απαραίτητο εξοπλισμό, όμω το πρόγραμμα αυτό καθεαυτό όπω έχει προταθεί δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει τέτοιο εξοπλισμό. Δεύτερη παρατήρηση. Και εδώ έχουμε μια επιφύλαξη για τι κατεξοδότηση πράξη. Η σχετική τροπολογία, όπω έχει κατατεθεί, μα οδηγεί στο εξή. Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα πρόγραμμα δοκιμαστικό για τα προγράμματα πληροφοριών και τις ανθρώπινες δραστηριότητες, δηλαδή κατάρτιση, σεμινάρια, εργαστήρια, που πρέπει να διοργανωθούν δεν έχει να κάνει με περαιτέρω δράσεις από τη στιγμή που θα εγκριθεί ο κανονισμός. Επίσης έχουμε επιφυλάξεις για μια άλλη κατηγορία για τις οροφές του προπολογισμού και τα σχετικά άρθρα στην ενδιάμεση αξιολόγηση. Τονίστηκε η ευελιξία του προγράμματος, μια από τις προτεραιότητες ε, του προγράμματος και ένα από τα βασικά του πλεονεκτήματα. Εάν λάβουμε υπόψη τις δυσχερείς οικονομικές συγκυρίες αυτή τη στιγμή και το γεγονός ότι δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί ενοποίηση των τελωνιακών υπηρεσιών στο 2020, νομίζω ότι με αυτά τα δεδομένα πρέπει να διατηρηθεί η ευελιξία του προγράμματος και να μπορεί να γίνει επανακατανομή των κονδυλίων ανάλογα με τις μεροντικές ανάγκες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας. Και το 0,25% του προπολογισμού ως οροφή γιατί διαχείριση του κόστου του προγράμματο είναι πραγματικά πολύ μικρό. Αυτό ήταν ένα σχόλιο ε, ε ίσονο σημασία επί των λεπτομεριών. Και τέλο, έχουμε κάποιε επιφυλάξει για την πρόταση που έχει να κάνει με του δείκτε. Δεν είναι σαφέ ποιοι είναι οι λόγοι ακριβώ που ο δείκτη αυτό προτείνεται από τον εισηγητή. Θα θέλαμε λοιπόν κάποιε ε, περαιτέρω εξηγήσει πριν προχωρήσουμε. Και εγώ ευχαριστώ. Θα ήθελα όμως αν μπορεί η Επιτροπή να απαντήσει στο ερώτημα του κυρίου Σμιτ όσον αφορά την συμμετοχή, την ενεργό συμμετοχή όσον αφορά τη χρηματοδότηση στα προγράμματα. Sorry, I didn't because he left. Ναι, δεν το απάντησε γιατί είχε φύγει. Ε, μπορεί κάποιο να του μεταφέρει την απάντηση. Ναι, υπήρξαν κάποια ερωτήματα από τον λόγο βουλευτέ. Πρώτα απ' όλα, ποια θα είναι η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων στο σύστημα. Πρέπει να σας πω ότι ετοιμάζουμε το πολιετές στρατηγικό πρόγραμμα μας, όπως το αποκαλούμε, το συζητούμε με τα κράτη-μέλη και θα το συμφωνήσουμε από κοινού με αυτά. Αυτό θα αποτελέσει τον οδικό χάρτη για την υλοποίηση όλων των υφιστάμενων ευρωπαϊκών συστημάτων πληροφοριών που χρηματοδοτούνταν ή μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το τελωνιακό πρόγραμμα μέχρι το 2013 ή από το επόμενο UCC. Είναι σημαντικό από πλευράς κομισιών και από πλευράς κρατών μελών να γνωρίζουν όλοι τι πρέπει να κάνουν και μέχρι πότε για να προγραμματίσουμε και τους προπολογισμού μας. Από πλευράς Κομισιών είναι προφανές ότι ο προϋπολογισμός θα προέρχεται μόνο από το πρόγραμμα του 2020, αλλά ε, στα κράτη-μέλη, κάθε κράτος καταρτίζει το δικό του προπολογισμό. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο ερώτημα, δηλαδή γιατί το σύστημα τα κενό μόνο για κάποια κράτη-μέλη. Ακούστε, αυτό οφείλεται στις ανάγκες που εντοπίσαμε και συγκεκριμένα. Εάν βάλουμε μαζί την προσπάθεια κάποιων κρατών μελών, είπαμε ότι αυτή η προσπάθεια μπορεί να ωφελήσει την όλη κοινότητα. Για παράδειγμα, μπορεί κάποια κράτη-μέλη να έχουν κοινέ ανάγκε ό,τι αφορά ένα συγκεκριμένο σύστημα, παραδείγματο χάρη τον έλεγχο των ισρώων. Και σήμερα γίνονται τα πράγματα 27 φορές. Μήπως θα ήταν καλύτερα κάποια κράτη-μέλη, 8, 9, 10, πρόθυμα, να δώσουν, ε, μάλλον να, να λάβουν κάποια δημοσιονομική στήριξη από το πρόγραμμα και μετά να παράγουν ένα αποτέλεσμα που θα είναι υποφελές για το σύνολο της κοινότητας. Έχουμε και το Expert Team που είναι ένα εργαλείο του νέου προγράμματος. Δεν θα γίνονται δηλαδή για όλα τα κράτη-μέλη κάποια πράγματα από την αρχή, αλλά για κάποια και μετά θα χρησιμοποιούν το αποτέλεσμα όλα τα υπόλοιπα. Κάποια σχόλια για τα μέτρα καταπολέμησης της απάτης, τη συνεργασία με την Όλαφ και ούτω καθεξής. Θέλω να σας ενημερώσω ότι πράγματι συνεργαζόμαστε στενά με την Όλαφ. Η Όλαφ χρησιμοποιεί το δίκτυο CCSCSA, e το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Τελωνία 2013 και είμαστε σε πολύ στενή επαφή μαζί με τον οργανισμό αυτό διότι χρησιμοποιεί όλες τις ευρωπαϊκές δομές που έχουμε για διασύνδεση όλων των κρατών μελών. Και αυτό χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Τελωνίου 2013 και γι' αυτό έχουμε και στην επαφή μαζί τους. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, λέει Νομίζω ότι προσθέσατε κάποια αξία στη συνόλη συζήτηση και θα δώσω τώρα το λόγο στον εισηγητή κύριο Παλτασάρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους, τον κύριο Σμιτ, τον κύριο Κοφεράτη, τον κύριο Μπίλαν, εσάς την ίδια, για τις ε, προτάσεις και τα επενδυτικά σχόλια που ακούστηκαν. Νομίζω ότι οι προτεραιότητες που τέθηκαν από τη χρηματοδότηση ως την ανάγκη να δοθεί έμφαση στην ασφάλεια, την καταπολέμηση της απάτη στο ρόλο των συστημάτων πληροφορικής είναι πραγματικά σημεία που βρίσκονται στην καρδιά του ενδιαφέροντός μας μαζί με τα υπόλοιπα που συζητήσαμε για το θέμα του προγράμματος αυτού. Αρκεί να σκεφτούμε τις απίστευτες ζημιές που λόγω της πειρατείας και της παραχάραξης ή της παραβίασης των προδιαγραφών για την επιστηστική ασφάλεια προκύπτουν στην ευρωπαϊκή οικονομία. Όλα αυτά περνούν από τα σύνορά μας. Βεβαίως δεν μπορεί κανείς να φανταστεί ότι το πρόγραμμα Customs για τα τελωνία δηλαδή θα εξασφαλίσει απόλυτη ασφάλεια, όμως είναι ένα συμπληρωματικό κριτήριο προτεραιότητας. Θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα λειτουργικό που να συμβάλλει αποτελεσματικά στην προστασία των συνόρων μας. Έτσι πρέπει να δούμε τα τελωνία. Με τη συλλογή πληροφοριών, τη συστηματικότητα συλλογής πληροφοριών, ως προς τα χρηματοδοτικά. Τα ποσοστά που προτείνουμε είναι τα ελάχιστα. Τα ελάχιστα που έχουν αποδοθεί στους διάφορους ε, τομείς. Τώρα, η ευελιξία είναι κάτι που επιθυμούμε να υπάρχει. Εύχομαι και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταλήξουμε σε συμβαστικά, συμβαστικές λύσεις που να φέρουν σε σύγκληση τις θέσεις των ΜΕΝ και των ΒΕ. Όμως θα πρέπει να υπάρχει μια αρχική διάκριση, βασική διάκριση των ποσών παρά να υπάρχει ασάφεια για τα διάφορα κεφάλαια του προγράμματος. Αυτό το θεωρήσαμε αναγκαίο. Ως τις 12 Νοεμβρίου μπορούν να υποβληθούν τροπολογίες, οπότε ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν στη συζήτηση για τη συνεισφορά τους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή τη συζήτηση. Ολοκληρώσαμε το θέμα αυτό. Θα ήθελα πραγματικά να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα το απόγευμα στις 3 θα ξεκινήσουμε με τον Επίτροπο Ταγιάννη. Ελπίζω να ενημερώσετε όλους τους συναδέλφους να είναι πολλοί συνάδελφοι παρόντες. Σήμερα το απόγευμα στις 3 παρακαλώ.